Is anyone from the Secretariat here? Okay. Right, ladies and gentlemen. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε τη σημερινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών. Θέμα πρώτο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αύριο βράδυ θα αλλάξουμε την συνεδρία των συντονιστών με την κυρία Χέλγκα Σμιτ και καθορισμό εισηγητή για την ε, αντιπροσωπεία για την Σερβία. Έχετε ήδη ειδοποιηθεί με email, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Λοιπόν, σημείο 2, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Και περνάμε τώρα στο σημείο 3 σύναψη της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΑΚ. Έχουμε λοιπόν πρώτη εξέταση του σχεδίου κοινή πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου για την σύναψη της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινική Αμερική και Καραϊβική με στόχο να ενισχυθεί η στρατηγική συνεργασία και η αυξημένη συμμετοχή τη κοινωνίας των πολιτών. Πέρυσι τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες Λατινικής Αμερική και Καραϊβική υπέγραψαν μια συμφωνία για το Διεθνές, Αυτοσίδρυμα, το Διεθνές Αυτοίδρυμα με και θα πρέπει να δώσει και την σύμφωνη γνώμη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δώσω λοιπόν τώρα τον λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Κούζο. τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το 1999 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική ξεκίνησαν μια διπεριφερειακή στρατηγική συνεργασία και το 2010 ε, κορυφώθηκε αυτό με τη σύσταση της ε, ΣΕΛΑΚ. Ε, το Ίδρυμα ιδρύθηκε και από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΛΑΚ το 2010 μαζί με την Ένωση αυτή ως ε, διακλάδωση ε, της ε, Ένωσης και προωθούν σχέδια στα πλαίσια της διαπεριφερειακής δράσης. Θέλουν να προωθήσουν λοιπόν αυτή την ε, διπεριφερειακή στρατηγική σχέση θεμελιώνοντας την ενεργό συμμετοχή και τις κοινωνίες των πολιτών και από τις δύο πλευρές υπάρχουν αρκετά προγράμματα τα οποία εξετάζουν αυτή τη περιφερειακή σχέση, ε, προωθούν ε, σημεία συνάντηση ε, για μη κυβερνητικού παράγοντε, ώστε να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε και να ενισχύσουμε την κυβερνητική διαδικασία για να δοθούν απαντήσει στι προκλήσει που αντιμετωπίζουν και οι δύο περιοχέ. Γίνεται ανάλυση και αναλύεται το θεματολόγιο ε, της διπεριφερειακής αυτής στρατηγικής συνεργασίας και υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις, έγγραφα, βιβλιογραφικές αναφορές κλπ. Το Ίδρυμα, κατά την άποψή μου, είναι πολύ σημαντικό παρακλάδι αυτής της Ένωσης, διότι ε, βοηθά σε κοινέ εργασίες για πολλά πράγματα κοινού ενδιαφέροντος. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις μέρες οργανώνεται ένα φόρουμ προβληματισμού για την οικονομική παραγωγικότητα και την ε, ε, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και το Ίδρυμα βοήθησε για να γίνει η επόμενη Πανεπιστημιακή Σύνοδος που θα περιλαμβάνει και την πλειοψηφία ε, του πανεπιστημιακού κόσμου των δύο περιοχών για να μπορέσουν να ξεχάσουν διαιρέσει και συγκρούσει που είχαν στο παρελθόν. Επίση, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να ε, ιδρυθεί αυτό το Ίδρυμα ω διεθνή οργανισμό για να μπορέσει να υπάρχει μια σχέση μεταξύ τη κοινωνία των πολιτών και τη Ένωση, η οποία θα εμπλουτίζεται από περισσότερα στοιχεία. Δυστυχώ υπήρχαν κάποια προβλήματα στη δράση του Ιδρύματο ε, επειδή ακριβώ ήταν ένα απλό ιδιωτικό Ίδρυμα. Πολλέ χώρες στα πλαίσια της ΕΛΕΚ δεν, το αναγνωρίζουν ως επίσημο ίδρυμα ε, παρά μόνο να αλλάξει νομικό καθεστώς και γίνει ένα διεθνές ίδρυμα. Έχει και συνέπειε για τη χρηματοδότηση βεβαίω του ιδρύματο αυτό και ελπίζουμε να είναι καλύτερα καταναμημένη μεταξύ των χωρών της ε, Λατινικής Αμερική και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το μεγαλύτερο βέρο τη χρηματοδότηση. Όπως είπαμε, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις αμοιβέ σχέσεις για να μπορέσουμε να έχουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους και τους Λατινοαμερικανούς πολίτες και να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες προκλήσεις. Επομένως, η κύρωση αυτού του Ιδρύματος ως Διεθνές Ίδρυμα είναι πλήρως αιτιολογημένη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. for your... ευχαριστούμε, συνάδελφε. προτείνω τώρα να δώσουμε τον λόγο στους κοιόδης εισηγητές, ε, όσοι είναι παρόντες. Αντώνιο Λόπες Εστούρες για το ΕΛΚΑ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μου ομάδα και εγώ συμφωνούμε με την ε, πρόταση του εισηγητή να ε, με αυτό το Ίδρυμα γιατί σίγουρα βοηθά τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών Λατινικής Αμερικής και ε, Καραϊβικής. Δίνουμε νομική προσωπικότητα σε αυτό το Ίδρυμα το οποίο από το 2010 κάνει πολύ σημαντική δουλειά για τη σχέση των χωρών αυτών. Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική ε, διπεριφερειακή σχέση η οποία δημιουργήθηκε το 1999 στην πρώτη σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινική Αμερικής ε, και Καραϊβικής ε, στο Ρίο Τζανέιρο ε, έδωσε πολλά στοιχεία και μπόρεσε να προωθήσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την πολιτική διάσταση και τη διεθνή συνεργασία βασιζόμενη σε σημαντικές εμπειρίες. Τα όσα έγιναν από τη στρατηγική αυτή ένωση ε, δείχνουν ευθύ εξ αρχή ε, ότι μπορούμε να έχουμε πολύ επιτυχημένε προσπάθειε και επομένω θα πρέπει να αλλάξει και το νομικό καθεστώ του Ιδρύματο για να μπορέσει να εργαστεί με πιο αυτόνομο και αποτελεσματικό τρόπο. Η ανάγκη να έχουμε ένα ίδρυμα διεθνού χαρακτήρα ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Περιλαμβάνονται και στην σύσταση της Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΑΚ και συζητήθηκε και στη Μαδρίτη και πιστεύω ότι όλα αυτά θα ενισχύσει και τις υπάρχουσες υποχρεώσεις των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του διπεριφερειακού διαλόγου και θα συνεισφέρει και θα μας βοηθήσει να καλύψουμε και τις προσδοκίες των Λατινοαμερικανών και των Ευρωπαίων πολιτών στην τελευταία σύνοδο στις Βρυξέλλες ε, ε, θέλαμε να έχουμε ε, κοινωνίες οι οποίες ευημερούν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και συμφωνώ με τον συντάκτη της έκθεσης ε, για το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι κάτι το οποίο μας αφορά και εμάς και υποβάλαμε και σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ασής είναι εδώ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ο κύριος Τάνοκ, ο κύριος Ασεβίτσιος, ο κύριος Καστάλτο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την κύρωση αυτή της συμφωνίας και φυσικά εκτιμώ και τα όσα εξήγησε ο εισηγητής προηγουμένως. Ε, το νομικό καθεστώς ε, είναι το επόμενο βήμα για αυτό το Ίδρυμα, το οποίο απέδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει ε, στη συνεργασία των κρατών ε, από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά είναι και θεμελιώδη σημασία για να μπορέσουν να έχουν και συνεργασία ε, οι κοινωνίες των πολιτών των αντίστοιχων χωρών. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι στην έκθεση, στη σχέση που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών Λατινική Αμερική και Καραϊβική, δεν θα πρέπει να τη βασίζουμε μόνο σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά πρέπει να είναι και σε πολιτιστικό επίπεδο με την ευρεία έννοια του όρου. Συμφωνούμε με τι ανησυχίε όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά συμφωνούμε απόλυτα και με τον εισηγητή ότι υπάρχει διάθεση να ακυρώσουμε τη συμφωνία και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα με μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση και ε, να υπερψηφίσουμε και όλοι εμείς εδώ στην Επιτροπή. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή για τη δουλειά του μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Καστάλντο. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Κύριε Κούσο, θα θέλατε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ναι, πολύ σύντομα. Απλώς ε, να χαρώ ιδιαίτερα για την ομοφωνία παρά το γεγονό ότι μόνο δύο σκιώδεις συγητές είχαμε εδώ αλλά χαίρομαι που για μια φορά συμφωνώ και με το ΕΛΚ και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να την μεταφράσουμε και σε κύρωση του Ιδρύματος αυτό, ε, να αλλάξει λοιπόν το νομικό της καθεστώς ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να θεμελιώνει αυτή την διπεριφερειακή συνεργασία. Τίποτα άλλο σας ευχαριστώ. Okay, thank you, dear colleague. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι στις 12 Ιουλίου, 11 η ώρα. Ωραία, λοιπόν. Περνάμε τώρα στο σημείο 4, στρατηγική ΕΕ Αφρικής, μια όθηση για την ανάπτυξη. Θα συζητήσουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης από τον κύριο Καστάλντο. Με την γνωμοδότησή μας θα συνεισφέρουμε σε μια έκθεση πρωτοβουλίας που προετοιμάζεται στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Η πέμπτη σύνοδος κορυφής Αφρικής ΕΕ θα πραγματοποιηθεί στο Αμπιτζάν στις 28 και 29 Νοεμβρίου και η έκθεση θα αποτελέσει μια συνεισφορά στην ε, συζήτηση πριν από την σύνοδο κορυφής. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Καστάλτο για να παρουσιάσει το σχέδιό του. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ε, πολύ σωστά υπενθυμίσατε και εσείς ε, και όπως συνειδητοποιούμε και όλοι, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Εσείς πολύ σωστά είπατε ότι 28 και 29 Νοεμβρίου θα γίνει αυτή η πέμπτη σύνοδος ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής που θα είναι ζωτική σημασία για την μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο υπήρων. Το 2018 θα ξεκινήσουν και διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μετά του Κοτονού, για να μπορέσουμε να έχουμε και μια πιο ε, καλά εδρωμένη ε, εταιρική σχέση με τις χώρες ε, αυτές. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το ψήφισμα. Εγώ είμαι και συντάκτης της γνωμοδότησης ε, εκ μέρους της Επιτροπής μας για να δώσουμε την κατάλληλη εντολή στους εκπροσώπους μας και να έχουμε και εκπεφρασμένες πολιτικές θέσεις της Επιτροπής μας. Η Αφρική τα τελευταία χρόνια σε πολύ βαθιές αλλαγέ και σε πολιτικό και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο και με τον ίδιο τρόπο, με τελείως όμως διαφορετικό τρόπο είχαμε αλλαγέ ε, και στην Ευρώπη. Ε, δεν μπορούμε να αναλύσουμε τις αλλαγές γιατί γίνονται στα πλαίσια ενός κόσμου ο οποίος είναι όλο ένα και πιο συνδεδεμένος και πιο σημαντικός. Υπάρχουν ε, υπερεθνικές προκλήσεις οι οποίες κατά την άποψή μου απαιτούν και μια κοινή προσέγγιση και είναι και πολλές. Ε, υπάρχει για παράδειγμα μια ολένα και πιο ασαφής παγκόσμια τάξη. Ε, η ασφάλεια, ο κίνδυνο τη τρομοκρατία, η αλλαγή του κλίματο και η μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι ο βασικό εταίρο τη Αφρική. Είμαστε οι πρώτοι στι ξένε επενδύσει και στι εμπορικέ συναλλαγέ. Είμαστε η πρώτη πηγή βοήθεια στην ανάπτυξη και φυσικά βοηθάμε και σε τομέα ασφαλεία. Ε, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και από πλευρά Αφρική βεβαίω υπάρχει κάθε ενδιαφέρον για να εμβαθύνουμε αυτή τη σχέση και υπάρχει φυσικά και η γνώση ότι αν δεν γίνει αυτό θα μα οδηγήσει και σε συνέπειε οι οποίε ε, επιτρέψε μου να πω και κατεφημισμό ότι θα είναι καταστροφικέ. Η ε, Επιτροπή το Μάιο του 2017 δημοσίευσε λοιπόν αυτή την κοινή ανακοίνωση για ανανέωση της ε, εταιρική σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής και εμείς ε, εκπονούμε τώρα αυτή την έκθεση. Εμείς ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πρέπει να γνωμοδοτήσουμε και να δώσουμε στην Επιτροπή Ανάπτυξη σε ένα κείμενο το οποίο θα καλύψει και τις προσδοκίες μας. Όπως γνωρίζετε το κείμενο πρέπει να είναι πολύ συνοπτικό αλλά είμαι βέβαιος ότι με την βοήθεια των σχεδόν εισηγητών και με τι τροπολογίε σα θα μπορέσουμε να το εμπλουτίσουμε περαιτέρω για να μπορέσουμε να εκφράσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τι προτεραιότητε μα και τι απόψει μα. Καταρχά ε, να πω ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική, όπω λέω και στην πρώτη παράγραφο και πρέπει να το βασίσουμε σε κοινά ενδιαφέροντα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι παγκόσμιες προκλήσει. Στην τρίτη παράγραφο που αναφέρομαι στην ασφάλεια επισημαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καλέσουμε του εταίρου μα να δημιουργήσουν ε, ευπροσάρμοστε κοινωνίε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην παιδεία και στις θέσει εργασία, ιδίως για τους νέους. Όπως εκδηγεί και η ανακοίνωση τη ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δημογραφική πρόκληση στην Αφρική είναι τόσο μεγάλη που θα φτάσουμε στα 2,4 δις ε, ε, μέχρι το 2050 στην Αφρική και ε, το 60% θα αποτελείται από νέους. Ε, γι' αυτό ακριβώ το λόγο πρέπει να δημιουργηθούν 18 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το χρόνο στην υποσαχάρη Αφρική για να μπορέσουμε να πάμε ε, στους ίδιους ρυθμούς με την ανάπτυξη του πληθυσμού. Είναι απίστευτη αυτή η πρόκληση αλλά και η πραγματικότητα είναι εξίσου απίστευτη. Εάν λοιπόν δεν μπορέσουν να πιστέψουν οι νέοι ότι έχουν αξιόπιστες δυνατότητε στη χώρα τους και θα μπορέσουν να ενταχθούν θα υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος περιθωριοποίησης κρίση, κοινωνικού αποκλεισμού που γνωρίζουμε και σήμερα μεταφράζονται σε μεταναστευτική πρόκληση και σε τρομοκρατία. Στην τέταρτη παράγραφο τονίζω ότι κάθε συνεργασία είναι επιθυμητή, αλλά ο τομέα τη ασφάλεια θα πρέπει πάντα να θεμελιώνεται στι βασικέ αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνάδει και με τι αρχέ τη δημοκρατία, τη πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των. Ε, ε, ίσων δικαιωμάτων. Τονίζω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα ε, αίτια της μετανάστευσης και θα πρέπει να υπάρξουν και συμπράξεις με τρίτες χώρες που δεν θα είναι απλώς σε ποσοτικό επίπεδο και σε έλεγχο των μεταναστών. Θα πρέπει να βασίζονται σε σοβαρό και συνεχή διάλογο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εταίρους μας σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο να αναπτυχθούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά μπόρεσα να έχω στην πρώτη εκδοχή του κειμένου. Ελπίζω να μπορέσω να συμπεριλάβω περαιτέρω τροπολογίε για να μπορέσω να καλύψω και αυτέ τι συγκεκριμένε συμμετοχέ. Περιμένω την συνεισφορά σα και είμαι ε, διατεθειμένο να συζητήσω και με του και ηγητέ για να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα περιλαμβάνει και του πάντε και θα είναι, ε, βρίσκει σύμφωνο στου πάντε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και του και ηγητέ ε, που είναι παρόντε στη συζήτηση. Βλέπω τον κύριο Τσέζα, τον κύριο Τζάρ, τον κύριο και τον κύριο Κούσο. Να σας πω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 12 Σεπτεμβρίου και ε, να πω ότι με μεγάλο ενδιαφέρον και με μεγάλο ενθουσιασμό περιμένω την συνεισφορά σας και τις, ε, τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Castaldo. Ευχαριστούμε κύριε Καστάλτο. Περνάμε τώρα στις δηλώσεις των σκιωδών συγητών. Λορέντσο Σέζα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Καστάλτο για την γνωμοδότησή του είναι συνοπτική μεν, αλλά περιέχει τα στοιχειώδη. Και πιστεύω ότι οι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική ε, γίνονται όλο και πιο σημαντικέ, και πρέπει να προσαρμόσουμε και τη στρατηγική μα για να ανταποκριθούμε στι παρούσε προκλήσει. Πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για να βοηθήσουμε την Αφρική να αντιμετωπίσει τι πολλέ προκλήσει που έχει, κυρίως οικονομική ανάπτυξη, αλλά τρομοκρατία και κλιματική αλλαγή επίση η συνεισφορία της Επιτροπής μας, ε, η οποία έχει σχέση και με τις βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάπτυξης, ε, δεν είναι απλώς ε, μία, ένα σχόλιο. Θα πρέπει να έχουμε μία συντονισμένη προσέγγιση σε θέματα μετανάστευσης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Πρέπει να πω ότι εκτίμησα ιδιαίτερα την αναφορά στο κείμενο στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Πά και ε, επίσης ε, στις ε, ευρωπαϊκές αποστολές, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες θα επιτρέψουν να έχουμε και σταθερότητα και είναι και η απαραίτητη βάση για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Από πλευρά ΣΕΛΚ νομίζω ότι θα υποβάλουμε περιορισμένε τροπολογίε, οι οποίε θα επικεντρωθούν κυρίω στι πολιτικέ πτυχέ τη συνεργασία μα για την Αφρική και μετά σε θέματα ασφαλεία και μετανάστευση. Ελπίζω και φαντάζομαι ότι το χρονοδιάγραμμα θα προχωρήσει γρήγορα και θα μπορέσουμε να είμαστε παρόντε ε, στο ραντεβού του Νοεμβρίου στην ακτή του Ελεφαντοστούν για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική. Thank Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον κύριο Ζάλ από τους Σοσιαλδημοκράτες. ευχαριστώ. Συνάδελφοι, να πω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης είναι ισορροπημένο, αλλά και αρκετά γενικόλογο και αποφεύγει τα δύσκολα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της ε, ΑΦΕΤ να φέρει μια πιο στρατηγική προοπτική στην συζήτηση αυτή. Κάτι το οποίο είναι επίγον δεδομένη της έκτασης ε, των αλλαγών στην Αφρική και των αντίκτυπο που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ευρώπη και για την εξωτερική μας δράση. Η Αφρική γίνεται στρατηγική προτεραιότητα εξίσου μεγάλη σημασία με την Ανατολική Γειτονία και τη Μέση Ανατολή. Και άρα θεωρώ ότι η Σύνοδος Κορυφής του φθινόπωρου θα είναι πράγματι κρίσιμη. Τώρα να συνεχίσουμε ο ε, συνήθως δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε νέες ιδέες και νέα όθηση. Ένα από τα βασικά στρατηγικά ζητήματα αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση και τους κινδύνους ενός νέου προστατευτισμού και τις ε, τάσεις αυτές στην Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε περισσότερο τα έργα αυτά, μεταξύ των οποίων και τις διάφορες συσσωματώσεις στην Ανατολική, Δυτική και Νότια Αφρική και να φροντίσουμε να συμπληρώνουν την παναφρικανική ολοκλήρωση που αντιπροσωπεύει η Αφρικανική Ένωση. Επίσης πρέπει να καλλιεργήσουμε διμερείς σχέσεις με τις χώρες Λιβιά την Νότια Αφρική, την Ιγυρία, την Αιθιοπία, που παίζουν ηγετικό ρόλο. Στην Βόρεια Αφρική πρέπει να αναζωογονήσουμε την Ένωση της Μεσογείου, που το ξεχάσαμε αυτό το αρκετά έξυπνο σχέδιο, για να ενθαρρύνουμε την κοινή ευθύνη για την περιφερειακή μας ασφάλεια. Ένα άλλο θέμα αφορά την Κίνα και τις στρατηγικές της επενδύσεις στην Αφρική. Είναι επιτακτική ανάγκη να έρθουμε σε επαφή με την ε, Κίνα ως εταίρο στην οικοδόμηση σταθερότητας και κράτους δικαίου στην Αφρική. Τέλος, θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάποια ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη την ε, διαφθορά που φτάνει σε βαθμό εχμαλώτισης του κρατικού μηχανισμού και τον μηχανισμό της ολιγα... του ολιγαρχικού πλουτισμού της κρατικής γραφειοκρατίας κάποιων αφρικανικών χωρών βεβαίω. Υπάρχει και το θέμα της τραγωδίας ε, των παράτυπων χρηματικών ροών, αλλά η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται αλλού. Γι' αυτό θα υποβάλω πολλές τροπολογίες και αναμένω βεβαίω μια επικοδομητική συζήτηση με τον κύριο Καστάλντο και με τον κύριο Πόγκα ίσως στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ζάλα. Το ECR δεν είναι εδώ. Άλτε λοιπόν, η κυρία Βάτμανς. Ευχαριστώ. Κύριε Σίτα. Θεωρώ ότι έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Συμφωνώ με τους δύο προλαλήσαντες συναδέλφους. Ε, θεωρώ ότι πραγματικά καταφέρατε να καταγράψετε κάποιες πολύ σημαντικές σκέψεις, μεταξύ των οποίων έχουμε πρώτα απ' όλα την πολιτική συνεργασία με την Αφρική και εδώ πέρα έχουμε βεβαίως δύο βασικά σημεία. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η μετανάστευση. Νομίζω πως όπως δείχνει και το τελευταίο ευρωβαρόμετρο, να δούμε το τι θέλουν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θέλουν να κάνει περισσότερα πράγματα η Ευρώπη για την ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Οπότε θα ήθελα να φανούν πολύ περισσότερο αυτά τα σημεία και θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Σωστά μιλάτε για τη συλλογική ασφάλεια και το θέμα της άμυνας και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Κάτι άλλο το οποίο νομίζω δεν έχει αναφερθεί αρκετά και θα κάνω κάποιες σχετικές προτάσεις που ελπίζω να τις στηρίξετε. Μιλάτε δικαίως για ευρωπαϊκές αξίες. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα δικαιώματα των γυναικών, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει στο θέμα αυτό στην Αφρική. Και τέλος, αν το θα γίνει με ε, έργα μικρής κλίμακας για να ενθαρρύνουμε τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην Αφρική. Γιατί μιλάμε εδώ πέρα για τον ρόλο των πρεσβειών, το τι μπορεί να κάνει ο ιδιωτικός τομέας το εμπόριο με την Αφρική, πράγματα τα οποία νομίζω μπορούν κάλλιστα να μας απασχολήσουν στην ΑΦΕΤ και τέλος βεβαίω πρέπει νομίζω να μιλήσουμε και για τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ερευνητών. Νομίζω πως ε, θα πρέπει να δώσουμε και εκεί βάρος για να είμαστε σωστοί εταίροι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην ΚΟΕ και ως Κόσο. Όχι. Η πράσινη λοιπόν. Όχι. Δεύτερος γύρος, λοιπόν, για το ΕΛΚΟ, κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι μιλάμε για τόσο σημαντικά ζητήματα όπως οι σχέσεις μας με την Λατινική, Καραϊβική και Αφρική. Υπάρχουν σημαντικά στρατηγικά θέματα εδώ. Παρά το ότι θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο ελιγμών όταν μιλάμε για την Αφρική. Σύμφωνο με την στρατηγική έμφαση που αποδίδει ο εισηγητής ε, και οι σκιώδες αλλά θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Θα ήθελα να προτείνω την διακοινοβουλευτική συνεργασία. Θεωρώ ότι στρατηγικά εστιάζουμε στην συνεργασία με την Αφρική και δικαίως επιλέξαμε δύο χώρες με τις οποίες έχουμε αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις, δηλαδή την Κένια και την Τανζανία. Οπότε υπάρχει κάποια βαθιά συνεργασία σε διακοινοβουλευτικό επίπεδο και μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό και οι συνάδελφοί μας, οι βουλευτές επίσης το ίδιο θεωρούν. Αν μιλήσουμε τώρα για ζητήματα πέρα από την ΑΚΕ, Αυτό είναι κάτι το θετικό. Και νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε τις ε, ευκαιρίες ε, βαθύτερης συνεργασίας. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Προσφάτως συζητήσαμε την σημασία του πολιτισμού στα διεθνή φόρα και νομίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε επιτυχώς διάφορες στρατηγικές και αυτό θα μας οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Όσον, μιλά, όσον αφορά τώρα τον πολιτισμό και τον διαπολιτισμικό διάλογο, θεωρώ πως και εδώ έχει πολλά να προσφέρει η Αφρική. Σας ευχαριστώ κύριε Πέτερλε. Ο κύριος Φρόιντ κατόπιν για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα μιλήσω αγγλικά. Α, έτσι μου ήρθε. Νομίζω, συμφωνούμε χωρίς να είμαστε εμπειρογνώμονες για την Αφρική, ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η Ήπειρος είναι η έλλειψη ενέργειας, ιδιαίτερα ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συνδυασμός ε, της θερμότητας της, του θερμού κλίματος συμβάλλουν σε αφόρητες ε, ε, συνθήκες διαβίωσης. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα για να ψήξουν τα σπίτια τους ή για να αντλήσουν νερό για να αρδεύσουν τα χωράφια τους. Αλλά υπάρχει μια λύση για όλα αυτά και λέγεται ε, ενέργεια εκτός του γενικού συστήματος. Δηλαδή, σε αντίθεση με τα δικά μας συστήματα που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στα νοικοκυριά, με την ενέργεια εκτός συστήματος μπορεί να ε, παράγεται ενέργεια μέσω ηλιακής ενέργειας. Υπάρχουν τέτοια έργα που χρηματοδοτούνται από αμερικάνικες εταιρείες κυρίως. Έχουν βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης σε απομακρυσμένα μέρη της Αφρικής σε μεγάλο βάθμο. Με ε, μπορούν με αυτόν τον τρόπο να φορτίζουν τα τηλέφωνα τους, να παρακολουθούν τηλεόραση και βέβαια να δροσίζουν τα ε, σπίτια τους και επίσης τα παιδιά τους μπορούν να κάνουν τα μαθήματά τους το βράδυ λόγω ε, του φωτισμού. Αυτές είναι θεραπείες που δεν ε, κοστίζουν μια περιουσία, αλλά που αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις βελτιώσεις που αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Με πολύ μικρά ποσά μπορούν να επιτευχθούν πάρα πολλά πράγματα και μπορούν να επιτευχθούν για τους ανθρώπους αυτούς που φεύγουν και έρχονται στην Ευρώπη τους, ε, τους στηρίζουμε, τους ε, ενσωματώνουμε βέβαια, αλλά αυτό θα στήχιζε πολύ περισσότερο παρά να τους βοηθάμε στη χώρα τους, στις χώρες τους. Ευχαριστώ κύριε Φρόιντ. Ο κύριος Νάτιν είναι ο επόμενος Συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν, αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο αφορά όλα τα υπόλοιπα. Εάν δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και εδώ αναφερόμαστε και στο πολιτικά ορθό από το νέφωμα μιας πραγματικότητας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που ξέρουμε εμείς, στη Μαυριτανία, στο Νίγηρα, στο Μάλι, στο Τσάντ, στο Σουδάν, στην Νότια Αφρική, στο Κονγκό, στην Ιγυρία, στο Καμερούν. Η ασφάλεια είναι ζωτική σημασία γιατί ο τζιχαντισμός και η τρομοκρατία είναι ουσιαστικό κομμάτι της χώρας. Το πρόβλημα είναι ότι η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, πάλιωσε και δεν ε, ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που φαινόντουσαν ότι δεν υπάρχουν, αλλά εμφανίζονται τώρα. Και αυτοί οι πληθυσμοί οι οποίοι ζητούν ανάπτυξη και ζητούν ένα καλύτερο κόσμο, το πρώτο που ζητάνε είναι να μην τους σκοτώνουν, να μην τους βιάζουν, να μην τους βασανίζουν και να μην πεθαίνουν λόγω του τζεχ... λόγω της τρομοκρατίας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτό το αγγελικά πλασμένο άρθρο 41, το οποίο δεν επιτρέπει ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, όταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι προτεραιότητα απαραίτητη για την ασφάλεια, για να μπορέσει να δημιουργήσει ασφάλεια ε, και να μπορέσει να κάνει ένα ξεκαθάρισμα της τσιχαντιστικής ε, τρομοκρατίας, θα πρέπει να υπάρχει στρατιωτική παρέμβαση. Και φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει λοιπόν να κάνει ε, μία επίκληση στην πραγματικότητα. Πρέπει να βγούμε από το πολιτικά ορθό, το οποίο είναι αυτοκτονικό, μειοπικό, ε, και αυτό ε, σημαίνει ότι δεν μπορεί να δράσει με στρατιωτικούς σκοπούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βγούμε από αυτό το εγκληματικό ε, ε, που γίνεται, να μην βοηθάμε τους αντάρτες ε, στο Μάλι όταν όπλα έχει ο τζιχαντιστικός στρατός, ο οποίος τους χρησιμοποιεί μεγάλη επιτελεσματικότητα. Πρέπει να προσγειωθούμε, να σταματήσουμε να πετάμε στα, στα σύννεφα, διότι θα λερώσουμε μεν τις αρβίλες μας, αλλά πραγματικά θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο με πραγματικό τρόπο και όχι με τα όσα λέει το άρθρο 41. Ευχαριστώ κύριε Νάρ. Το τελευταίο ομιλητή είναι ο James Χαβ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω ε, και μπορούμε να καθίσουμε με τον κύριο Μπαστάλτο με τροπολογίες που θα ετοιμάσω. Θέλω να δούμε τα πράγματα από την κοινή λογική. Ε, με όλο το σεβασμό προς τον κύριο Ζάλα ανησύχησα που είπατε ότι πρέπει να στηριχθούμε στην Κίνα σε σχέση με τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Νομίζω αυτό γύρει ανησυχίες. Θα πρέπει να είναι καλό ότι αναφέρεται σε μια ισχυρή βάση Ηνωμένων Εθνών. Ε, θα πρέπει να δούμε ε, συνεργασία με άλλους οργανισμούς επίσης και ε, δεν μπορούμε να έχουμε μία λύση για όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα που αφορούν πολύ, πολύ συγκεκριμένες περιοχές της Αφρικής, πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει ξηρασία, λειψιδρία στην Ήπειρο. Θα υπάρξουν κάποιες τροπολογίες και σε αυτό το ζήτημα επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χάβερ. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Κάποιος άλλος από τους συναδέλφους. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τάσο Βινταλόγκα το, από την ΕΙΕΔ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε το σχέδιο ε, έκθεσης του κύριου Πόγκο και του κύριου Καστάλδο την, ε, το σχέδιο Τα Καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα θέματα του κοινού ανακαινθέντος από την Επιτροπή με μια επικοδομητική προσέγγιση και εκτιμούμε την σημασία που αποδίδεται στις συνιστώσεις ε, και τις διάφορες, ε, ε, τα διάφορα θέματα όπως είναι και ασφάλεια, εμπόριο, ανθεκτικότητα, θέματα που αφορούν την ενέργεια, και ευρύτερη συνεργασία. Θέλαμε να, μάλλον, να τονίσουμε την σημασία της κοινοβουλευτική συμμετοχής σε αυτή την συνεργασία, προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής. Ε, η χρονική στιγμή αυτής της έκθεσης, ε, εάν πετύχει, θα είναι ακριβώς πριν από τη Σύνοδο Κορυφής και υπάρχει και μια διακοινοβουλευτική συνάντηση του Ευρωκοινοβουλίου με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφή. Θα, ένα σχόλιο ουσία σε αυτό το στάδιο ε, θα είναι μια σύσταση ε, σχετικά με τον τίτλο της έκθεσης. Αναρωτιόμαστε ε, και που αναφέρεται στρατηγική υψηλόπιου Αφρικής, μια όθηση για την ανάπτυξη, αν θα μπορούμε να το πούμε ε, εταιρική σχέση ΕΕ Αφρικής, διότι υπάρχει μια κοινή στρατηγική ΕΕ Αφρικής, υπάρχει ε, ιδέα αναθεώρησης αυτής της στρατηγικής, αλλά θέλουμε να δώσουμε έμφαση στη σημασία ε, του, ότι αυτή είναι μια κοινή στρατηγική και αν έχουμε ένα ε, έντυπο που αναφέρεται στη στρατηγική ΕΕ Αφρικής, δίνει την εντύπωση ότι εμείς ορίζουμε μια μονομερή στρατηγική από δική μας πλευράς. Αν μπορείτε να εξετάσετε ε, μια αναδιατύπωση ε, ή να αναφέρετε στην κοινή στρατηγική ΕΕ Αφρικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα αίτημα ομιλίας ε, από την Κομισιόν, κύριος Ντομίνικο Ρόζα, επικεφαλής της μονάδας της Digitefco. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση και νομίζω πως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η γνωμοδότηση της Επιτροπής σας. Θεωρώ πως υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα πρέπει να τονιστούν. Πρώτα απ' όλα να έχουμε την γεωπολιτική σημασία της συνόδου αυτής θεωρώ πως έρχεται σε μια στιγμή όταν οι παγκοσμίες ισορροπίες αλλάζουν και αυτό έχει μεγάλη σημασία και πολιτική για το μέλλον. Δεύτερον, το ότι θεωρώ ότι σε κάποια σημεία της έκθεσης πρέπει να τονίσουμε το ότι η Αφρικα είναι και θα παραμείνει ο σημαντικότερος πολιτικός μας εταίρος. Είναι η κοντινότερη ήπειρος σε εμάς, με πολλές κοινέ προκλήσεις. Οπότε είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε σε έναν βαθμό. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι υπάρχει τίτλος για αυτήν την σύνοδο κορυφής που λέγεται «Επενδύουμε στην νεολαία». και βεβαίως ε, δούμε ότι τίτλος ε, φέτος ήταν για την Αφρική το πώς θα εκμεταλλευτούμε θα εκμεταλλευτούν ε, το δημογραφικό μέρισμα μέσω της ανάπτυξης. Και τέλος, τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πρέπει να υπάρχει κάποια στήριξη για να μπορέσουμε να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής ε, με μία φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Θεωρώ πως η ανακοίνωση της Άνοιξης τόνισε έξι προτεραιότητες ε, που νομίζω αναγνωρίζονται λίγο πολύ στην έκθεση αλλά θα μπορούσε να γίνει και μία πιο συγκεκριμένη αναφορά. Ξανά τέλος, οπωσδήποτε, ίσως ξέρετε πως ο τίτλος ε, θα είναι σύνοδος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ένωση, τώρα που αποφάσισε να ενταχθεί και το Μαρόκο. Κάτι το οποίο βεβαίως ε, θα πρέπει να έχει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο. Κύριε Καστάλτο, μια τελευταία παρατήρηση βεβαίως. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις μόνο για να απαντήσω και στα όσα ανέφεραν οι συνάδελφοι. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, η οποία ε, μου έδωσε πάρα πολλές ε, απόψεις. Θα μπορούσα να πω ε, ότι 1500 χαρακτήρες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμπεριλάβουν όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν. Ίσως θα χρειαζόμασταν τα δεκαπλάσια. Αλλά ε, ελπίζω με τη βοήθειά σας και τη συνεισφορά σας να μπορέσω να εμπλουτίσω περαιτέρω το κείμενο και να το διευρύνω. Όσον αφορά την άποψη του κυρίου Τσέζα για την ασφάλεια για μας προφανώ αποτελεί προτεραιότητα και όπως είδατε αφιερώσαμε και ειδική παράγραφο για το θέμα αυτό. Ε, σκοπεύουμε να το διευρύνουμε περισσότερο χωρίς όμως να ε, ε, έχουμε και ένα όρομα καθαρά στρατιωτικό γιατί εμείς θα θέλαμε το στοιχείο της ασφάλειας να περιλαμβάνεται με μια πιο ευρεία έννοια και να θεμελιώνεται στην ανάπτυξη ε, και στην εξέλιξη, να μην είναι σε στάσιμο επίπεδο, αλλά να υπάρχει ε, ένα σφαιρικό όραμα για να μπορέσουμε να επισημάνουμε τις βασικές πτυχές, χωρίς να πρέπει να επικεντρωθούμε απλώς και μόνο σε μία. Σίγουρα θα το επεξεργαστούμε περαιτέρω. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του κυρίου Τζάλα, ε, συμφωνώ με την ανάγκη να επεκτείνουμε περαιτέρω το στρατηγικό στοιχείο στη γνωμοδότηση αυτή. Ε, βέβαια θα μπορούσα εδώ να πω ότι παρά το γεγονό ότι αντιλαμβάνομαι την άποψή σα για τον προστατευτισμό, ε, αναλύοντας όμως την κατάσταση που έχουμε σε αρκετέ ε, περιοχέ τη Υπήρου, ε, για παράδειγμα ε, την κατάσταση στι μεγάλε λίμνε, αυτή τη στιγμή, αντί για τον προστατευτισμό θα έπρεπε να σκεφτούμε κάτι πιο θεμελιώδε. την προστασία για παράδειγμα. Υπάρχουν ολόκληροι λαοί, όπω για παράδειγμα ο λαό του Μπουρούντι, για τον οποίο είχαμε και κατεπήγον ψήφισμα στην τελευταία συζήτηση στο Στρασβούργο, που ε, κινδυνεύει με γενοκτονία. Ε, και φυσικά συμφωνώ απόλυτα, νομίζω ότι το είπανε και αρκετοί από τους ομιλητές, ότι πρέπει να ε, σταθούμε στην περιφερειακή συνεργασία, δηλαδή την παναφρικανική συνεργασία, αλλά και τη διμερή συνεργασία, δηλαδή να εδραιώσουμε κάποιες σχέσεις με κάποιες χώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να προσελκύσουν και τις υπόλοιπες χώρες της Υπήρου. Και πιστεύω ότι το θέμα των κινέζικων οικονομικών επενδύσεων θα πρέπει σίγουρα να το εξετάσουμε φτάσουμε, διότι πλέον η Κίνα, ε, επειδή έχει και το γεωπολιτικό αλλά και το οικονομικό διαμέτρημα το οποίο μπορεί να της επιτρέψει πλέον να γίνει παγκόσμιος παράγων και να έχει παρουσία παντού, έχω προσωπικά πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Δεν ξέρω αν ήταν και λάθος στη μετάφραση, ε, αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας ε, με την Κίνα. Σίγουρα θα είναι περίπλοκη αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα θα πρέπει να την αναλύσουμε αυτή την πτυχή, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ και την εσωτερική πολιτική πολλών αφρικανικών χωρών. Όσον αφορά τώρα τα όσα είπε η κυρία Βάουτμανς ε, για τις ευρωπαϊκές αξίες, ε, ναι, αναφερθήκαμε εντάχει στη σημασία της παρουσίας των γυναικών ε, στην ε, αστική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της Αφρικανικής Υπήρου και σίγουρα συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να διευρύνουμε περαιτέρω και να εμβαθύνουμε αυτή τη σχέση. Θα υπάρχουν όμως ε, δυνατότητες να το κάνουμε, όπως επίσης πιστεύω ότι και ο πολιτιστικός τομέας είναι αποφασιστική σημασίας και θα πρέπει να προωθήσουμε ε, συμπράξεις, ενεργασίες ε, και ίσως και προσχώρηση αφροκανικών χωρών σε ήδη υφιστάμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε ο πολιτισμός και η παιδεία να γίνουν καθολικό ε, προνόμιο και να μην είναι απλώς ε, προνόμιο ε, για λίγες χώρες. Και όπως είπε και ο κύριος Πέτερλε, αλλά το ακούσαμε και στις παρεμβάσεις του εκπροσώπου της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Κομισιόν, είναι πάρα πολύ σημαντική η διακοινοβουλευτική συνεργασία και πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής θα πρέπει ε, να είναι στο ίδιο επίπεδο ε, και χωρίς να θέλουμε να διδάξουμε εμείς τους εταίρους μας ή να τους επιβάλλουμε τι να κάνουμε. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι δεν μπορούμε εμείς ως, ως Επιτροπή, ε, γιατί απλώς μια γνωμοδότηση εκφράζουμε να αλλάξουμε το όνομα της σχέσης. Αυτό θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Αλλά φυσικά είναι μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να γίνει στην Επιτροπή ΔΕΒΕ. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ακόμα και αυτά που είπε ο κύριος Φρόιντ ε, για την ε, ενεργειακή πρόκληση και την ε, πρόκληση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά όπως το νερό. Σίγουρα δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Εσείς αναφέρατε και κάποια διαδεδομένα προγράμματα τα οποία απέδειξαν σύν το χρόνο ότι βοηθούν και έχουν μια εξαιρετική σχέση κόστους-οφελίας γιατί δημιουργούν και κάποιες εταιρικές σχέσεις πολύ καλύτερε παρά το γεγονό ότι είναι και πιο δαπανηρέ. Δεν ξέρω βέβαια πώ θα μπορέσουμε να τι εκμεταλλευτούμε και δεν ξέρω ε, αν αυτό είναι και αρμοδιότητα τη Επιτροπή ΔΕΒΕ. Αλλά πιστεύω ότι και εμεί θα πρέπει να εκφράσουμε την υποστήριξη τη Επιτροπή μα σε αυτή την προσέγγιση, σε αυτό το όραμα στην ε, ανάπτυξη και να υπάρχει και προσαρμοστικότητα για την Ήπειρο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς ε, για τις πολύ χρήσιμες παρεμβάσεις ε, και για τη σημασία που προσδώσατε ε, στην πρότασή μας ε, και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση που θα είναι ε, έργο όλων και θα επικεντρώνεται στην αμοιβαία συνεργασία, ίσης, επί ίσης με τις δύο υπήρους, αλλά να δώσουμε και βοήθεια στα 2 εκατομμύρια νέων ε, της Αφρικής που βλέπουν πλέον όλο και πιο αβέβαιο μόλον και σχεδόν χάνουν κάθε ελπίδα. Από αυτή την εταιρική σχέση μπορεί να γεννηθεί και η δυνατότητά μα να τους δώσουμε απαντήσει, να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των χωρών, μας, των χωρών τους και η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωση Αφρικής να μην είναι μονομερής, αλλά να είναι μια ισορροπημένη σχέση που θα βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό και ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Καστάρδο. Υπάρχει κανεί άλλο που θέλει να μιλήσει όχι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι είχαμε μια συνάντηση στο φορμά 5 συν 5 την περασμένη εβδομάδα. Σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι ήταν οι πέντε πρόεδροι των επιτροπών ε, με τους πέντε επιτρόπους που ασχολούνται με θέματα εξωτερικών υποθέσεων. Συζητήσαμε το θέμα αυτό και ε, συμφωνήσαμε ότι θα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα όχι μόνο για το 2017 αλλά και τα επόμενα χρόνια που ακολουθούν. Θα ε, γίνει ε, μια ε, ε προπαρασκευαστική συνάντηση πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στις 27 και 28 έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτοί που ενδιαφέρονται να παρευρεθούν σε αυτή την προπαρασκευαστική κοινοβουλευτική συνάντηση πρώτη συνόδου ε, θα έχετε ε, προσέξει ότι η καγκελάριος Μέρκελ ζήτησε ένα σχέδιο Marshall τίποτα λιγότερο από ένα σχέδιο Marshall για την Αφρική την περασμένη εβδομάδα. Είναι μέρος ε, της ατζέντα, βέβαια, της προεκλογικής ατζέντα στην Γερμανία. Αυτή είναι μια σημαντική έκθεση. Το χρονοδιάγραμμα έχει ω εξή. Η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι στι 13 Ιουλίου, στι 11 το πρωί, σε τρει μέρε. Η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα γίνει στις 30 ή 31 Αυγούστου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΔΕΒΕΣ 9-10 Οκτωβρίου. Είμαστε λίγο πολύ στην ώρα μας. Έχουμε φτάσει στο επόμενο σημείο. Ε, πρόκειται για δημόσια ακρόαση για το ρόλο των μελλοντικών συνολικών συμφωνιών με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Θα ήθελα να, καλωσορίσω, να σας καλωσορίσω σε αυτή την ακρόαση για τις μελλοντικές συμφωνίες. Οι ομιλητές παρακαλώ να καθίσουν εδώ ε, στο Προεδρείο και ε, μπορείτε να προσέλθετε εδώ στο Προεδρείο. So, ladies. Καλώς ορίζω την κυρία Μίνα Σιάν και την κυρία Αλιέβα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνάδελφοι, εισαγωγικά θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αναδιαμορφώνει τη σχέση της με την Αρμενία και με το Αζερβαϊτζάν μέσα από νέες συμφωνίες για τις οποίες οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν στην αρχή του χρόνου για την Αρμενία ή μόλις ξεκίνησαν στην περίπτωση του Αζερβαϊτζάν. Και στις δύο περιπτώσεις η Επιτροπή μας θα προετοιμάσει εκθέσεις, μια διαδικασία έγκρισης για την Συμφωνία ΕΕ Αρμενίας και μια ενδιάμεση έκθεση με συστάσεις προς τους διαπραγματευτές για την Συμφωνία ΕΕ Αζερβαϊτζάν. Η Επιτροπή ήδη πραγματοποιήσει μια επίσω αποστολή στην περιφέρεια πριν από δύο μήνες για να εξοικειωθεί με τα θέματα ε, στην περιοχή. Σήμερα έχουμε μια ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων με δύο εμπειρογνώμονε εν ώψη των, ε, της των δύο εκθέσεών μα. Οι δύο συμφωνίε αναμένονται να είναι συνολικές, τόσο στον αριθμό των θεμάτων που θα καλύψουν, όσο και στο βάθος τους. Οι ευκαιρίες και το κόστος αυτών των νέων σχέσεων και για την υψηλοεψηλό και για τους εταίρους είναι το πρώτο θέμα το οποίο χρειάζεται να ελέγξει το Κοινοβούλιο. Αυτές οι συμφωνίες αποτελούν ευκαιρία να ε, δώσουμε μια όθηση στην πρόοδο στην περιοχή για τις κύριες αξίες, δημοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση, κράτος δικαίου, ε, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χωρίς ε, καταπολέμηση της ε, διαφθοράς, μιας βαθύτερης οικονομικής συνεργασίας, αυτά παραμένουν μόνο νεκρό γράμμα. Τέλος, οι συμφωνίες έχουν, διατρέχουν τον κίνδυνο να υπονομευθούν από εξωγενείς παράγοντες, όπως περιφερειακές συγκρούσεις ή ξένες παρεμβάσεις, όπως έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Αναμένουμε από τους εμπειρογνώμονες να μας ρίξουν φως σε αυτά τα κέρια θέματα και να εισηγηθούν ε, συστάσεις πολιτικής ε, τις οποίες θα εξετάσουμε όταν επεξεργοζόμαστε τις εκθέσεις μας. Έχουμε καλέσει εδώ δύο ε, γνωστούς εμπειρογνώμονες για να παρουσιάσουν τις γνώμες τους επί των θεμάτων και εκπροσώπους από την ΕΕ που θα βρίσκονται μαζί μας σύντομα. Ο αρχικός ε, ομιλητός μας ήταν, ο ομιλητής μας ήταν ο κύριος Ρίσαρ Κυρακοσιάν, ο οποίος ε, λόγω κάποιου θέματος υγείας ε, δεν βρίσκεται μαζί μας. Έχουμε την κυρία Μίνα που είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Open, Foundation, Open Society Foundation της Αρμενίας έχει ε, εργαστεί για αυτό το Ίδρυμα εδώ και 19 χρόνια, υποβοηθώντας τις ε, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και προωθήσει των αξιών όπως κράτος δικαίου, ε, δημοκρατικές εκλογές, σεβασμός των μειονοτήτων και μια όθηση στην κοινωνία των πολιτών. Επίσης, κυρία Αλιέβα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και είναι η ιδρύτρια του Κέντρου Εθνικών και Διεθνών Σπουδών ενός, μιας δεξαμενής σκέψης που βρίσκεται στον Πακού του Αρτζερμπαϊτζάν. Προηγουμένως εργάστηκε και για ε, το ΝΑΤΟ, το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, ε, το Ινστιτούτο ε, Ανοιχτής Κοινωνίας και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. αναμένουμε γύρω στις 4.30 και τον κύριο Ντέρκ Σούμπελ από την ΕΕΣ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο ε, στις ομιλήτριές μας. Κυρία Μινασιάνη, κυρία Λιέβα, έχετε το λόγο. Thank you. Σας ευχαριστώ, κύριε Μακάλιστερ. Και καλησπέρα σας. τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που έχω να σας μιλήσω σήμερα, αν και όχι για τόσο ευχαριστώ λόγο, καθώς ο Ρίτσαρντ δεν μπορούσε να έρθει να εκφωνεί στην ομιλία του. Θα ξεκινήσω με την εμπειρία μου από τα Open Society Foundations και το πώς συνεργαζόμαστε με το Σύμβουλο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αρμενία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ορθή διοίκηση, τη χρηστή διοίκηση και το κάτω Έχουμε λοιπόν κοινωνία των πολιτών, μια συνάφεια θα έλεγα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια μεταρρυθμιστική ατζέντα η οποία έχει από κοινού με την Ευρώπη χαραχθεί ως η βασική κινητήριος δύναμη προς μια πιο ανοιχτή κοινωνία που θα κυβερνάται ε, καλύτερα και πιο δημοκρατικά. Γι' αυτό ακριβώς ε, προωθούμε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκινώντας με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, αλλά και πριν από αυτό, όταν είχε ενταχθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης Ερμηνεία και έτσι προσπαθούμε να παρακολουθούμε προσεκτικά το πώς είχε σχεδιαστεί η μεταρρύθμιση και προσπαθούμε να θέσουμε τα ζητήματα της χρηστής διοίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της λογοδοσίας σε πρώτο πλάνο και προσπαθούμε ακριβώς το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρούν αυτές τις υποσχέσεις. Και η προοπτική υπογραφής ε, της Συμφωνίας ε, Πλαίσιο ε, βεβαίως είναι κάτι το οποίο η κοινωνία των πολιτών στην Αρμενία και η ευρύτερη κοινωνία βλέπει πολύ θετικά. Αν δείτε τις έρευνες θα δείτε πως πάντα η επαφή με την Ευρώπη ήταν κάτι το οποίο έβλεπαν πολύ θετικά οι άνθρωποι στη χώρα και εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτή την ευκαιρία μετά από τέσσερα χρόνια, σχεδόν τέσσερα ολόκληρα χρόνια από το Σεπτέμβριο του 2013 όταν ελήφθη η απόφαση να μην υπογραφεί μόνο μερός ε, από την Αρμενία η Συμφωνία Σύνδεσης και είδαμε βεβαίως κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν ε, το τι σημαίνει αυτό για ολόκληρη την ε, κοινωνία της Αρμενίας. Για τον λόγο αυτόν καλωσορίζουμε την ευκαιρία αυτή για μια δομημένη και δεσμευτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και Για να ξεκινήσω τώρα, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω ποια είναι η κατάσταση και το τι έγινε τα τελευταία αυτά τέσσερα χρόνια. Η Αρμενία προσφάτως τον Απρίλιο είχε τις πρώτες βουλευτικές εκλογές με το νέο σύνταγμα. που στόχο έχει τη μετάβαση της χώρας από μια προεδρική σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οπότε ξεκινάμε τώρα σε ένα χρονοδιάγραμμα ενός έτους όπου θα ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση και ακριβώς πριν από τις εκλογές είχαμε την μονογραφία αυτή της συμφωνία πλαίσιο και από τι δύο πλευρές. Οπότε, οι εκλογέ αυτές ε, αποτέλεσαν την αρχή μια νέας περίοδου στην ζωή της χώρας ε, ως μια περίοδο μεταβατική. Γιατί έτσι ξεκίνησαν οι αλλαγές, ε, που προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας. Δηλαδή θα έχουμε σοβαρές νομοθετικές αλλαγές για το ποινικό δίκαιο, για τη χρηστή διοίκηση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έτσι έχουμε πραγματικές ευκαιρίες να αλλάξει η χώρα και να γίνει αυτό το οποίο ακριβώς ε, δηλώνει ως στόχο το Σύνταγμα. Δηλαδή να παρέχει καλύτερη διοίκηση, ε, ικανότερη δικαιοσύνη, διαχωρισμό των εξουσιών και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλες αυτές είναι αλλαγές που αφορούν άμεσα αυτούς τους τομείς της διοίκησης και της δικαιοσύνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έχοντας λοιπόν αυτό κατά νου, θα πρέπει πάντα να ερμηνεύεται αυτήν την περίοδο. Το δεύτερο είναι η πολύ αρνητική ερμηνεία, ε, με συγχωρείτε εμπειρία, της μη υπογραφής ε, της συμφωνίας του 2013 και προσπαθούμε να μάθουμε όσο περισσότερα μπορούμε από αυτήν την περίοδο έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο ή για να τα δούμε θετικά το πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως την περίοδο πρώτης υπογραφής. Το τι μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή και το τι πρέπει να μας απασχολήσει. Και θα ήθελα να πω πως ε, δυστυχώς ε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μας ανησυχούν και μας κάνουν επιφλεκτικούς. γιατί τα τελευταία τέσσερα χρόνια ή και πιο πριν είχαμε σοβαρές ε, οπισθοχωρήσεις στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ε, διοίκησης της χώρας είχαμε μια κατάσταση όπου οι πολιτικές ε, διαμαρτυρίες, η πολιτική διαφωνία και ακόμα και ο ακτιβισμός ε, υφίσταται πιέσεις. Ο κόσμος δεν έχει την δυνατότητα ή έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες να προσφύγει στα δικαστήρια λόγω του ότι είναι εξαρτημένη η δικαιοσύνη. και θα έλεγα ότι έχει φτάσει η στιγμή δεδομένων των μεγάλων νομοθετικών αλλαγών ακριβώς ε, να προσέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ζητήματα αυτά. Επίσης ε, πρέπει να θυμόμαστε ότι μετά τις εκλογές ε, του Απριλίου υπάρχει σοβαρή κοινωνική και οικονομική και μάλλον πολιτική άλλαγη, μάλλον κάποιες προετοιμασίες που γίνονται στη χώρα. Και συγκεκριμένα, όπως έχουμε πει, έχουμε συγκεντρωτική πολιτική εξουσία γύρω από τον πρόεδρο στην Αρμενία. Και τώρα για να έχουμε μια μετάβαση σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα υπάρχει η πρόκληση ε, σε ένα μέρος του καθεστώτος του πώς θα μπορέσει να διαχυθεί η συγκεντρωτική εξουσία σε ένα νέο σύστημα χωρίς να την χάσουν ουσιαστικά προσθέχουν δηλαδή τον ίδιο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας και της δικαστικής ε, και του Κοινοβουλίου στο νέο σύστημα. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ λοιπόν και να προβλέψουμε τα πράγματα αυτά στις νομοθετικές αλλαγές, να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να είναι ελεύθερος ο δημόσιος χώρος από την εξουσία αυτή που είναι τώρα συγκεντρωμένη γύρω από τον πρόεδρο. Και ένας τρόπος ε, να γίνει αυτό είναι να προσέχουμε τις αλλαγές που γίνονται από το νέο πρόγραμμα που λέγεται Ένωση Στρατού και Λαού όπου υπάρχει η πιθανότητα στρατιωτικοποίησης ε, της ε, κοινωνίας ε, και ευρέωσης κάποιων λειτουργιών της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένες συστάσεις που θα έκανα είναι η εξή. Θα πρέπει να δούμε τις μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης και να προσέξουμε ακριβώς ε, το θέμα του ποινικού κώδικα, του κώδικα ποινικής δικονομίας, να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει προτεραιότητα στον τομέα του ποινικού δικαίου και έχει επενδύσει πάρα πολλά εκεί. για να υπάρχει πρόληψη και δίωξη και καταστολή των βασανιστήριων. Αυτό είναι ένας τομέας όπου έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες και Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε ιδιαίτερως ε, τις μεταρρυθμίσεις ε, στον τομέα αυτών ε, όπως εξελίσσονται. Υπάρχουν κάποια θέματα στην κοινωνία στα οποία γίνεται μία κατάχρηση για να Υπάρχει μία αρνητική αντιμετώπιση της Ευρώπης, ε, ειδικά τα ζητήματα της οικογενειακής βίας, ε, της κατάργησης των διακρίσεων, των αντιδιακρίσεων. Αυτά θα πρέπει να τα προσέξετε πάρα πολύ. και να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις ε, της κοινωνίας ε, των πολιτών τα τελευταία χρόνια, όπως είπα. Ε, είχαμε αρνητικές εξελίξεις στην συμμετοχή του κοινού στην ελευθερία της έκφρασης, στην δυνατότητα έκφρασης αντίθετης γνώμης, και στο δικαίωμα του συνέρχεστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δικάζονται για πολιτικές απόψεις, πολιτικές φιλοδοξίες, επειδή είχαν άλλη άποψη από το κυβερνόν κόμμα και η πρόσβαση στην δικαιοσύνη των ανθρώπων αυτών είναι πολύ περιορισμένη και αυτή είναι τομής όπου ελπίζουμε να δώσει βάρος η Ευρωπαϊκή Ένωση και να φανεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέρος, ως συνομιλητής που θα επιμένει στα θέματα μιας ένωσης που βασίζεται σε αξίες. αντί απλά να είναι ένα συμβαλόμενο μέρος. Η εμπειρία που είχαμε με τις μεταρρυθμίσεις ε, στην Αρμενία δεν ήταν ικανοποιητική την έννοια ότι είδαμε μια επιφανειακή προσέγγιση στην μεταρρύθμιση και όχι πάντα επαρκείς απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιες συμπεριφορές. Δυστυχώς αυτό συνέβαινε πριν να ξεκινήσει η συμφωνία σύνδεσης και δυστυχώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ίδια αντιμετώπιση αλλά και κάποιες ε, εικασίες ε, για ζητήματα που είναι στην ημερήσια διάταξη ή είναι προτεραιότητες της Ένωσης. Και αυτό βεβαίως μας ανησυχεί. Και, όπως ε, προσπάθησα να πω, αυτά είναι θέματα που αφορούν ειδικά την προστασία του δημοσίου χώρου, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεστε, της αντιδιακρίσεις ε, και την οικογενειακή βία. Αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία θα δίναμε βάρος αλλά ιδιαίτερα οι τομείς ε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παίξει σημαντικό ρόλο στο να προωθήσει την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ορθή διοίκηση και την θέση που εκφράζεται τώρα από την τοπική αντιπροσωπεία εκεί. Είναι πολύ σημαντικό προσερχόμενοι στις ε, διαπραγματεύσεις να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το τι δεν πήγε καλά και να αποφύγουμε το να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και εδώ οι, διαπραγμα... διαπραγματεύσεις και η λογική του να ζητάμε λογοδοσία από τους Αρμένιους εταίρους μας έχει μεγάλη σημασία. Γιατί έχουμε δει κάποια επιδείνωση της κατάστασης και αυτό μας υπενθυμίζει την κατάσταση που υπήρχε Ειδικά όταν μιλάμε για την δικαιοσύνη και όταν μιλάμε για την οπισθοχώρηση της δημοκρατίας. Το θέμα είναι λοιπόν το εξής. Ενώ διαπραγματευόμαστε την συμφωνία και τσακάρουμε κουτάκια, ε, από φαίνεται θεωρητικά γίνεται πρόοδος, πρέπει να δούμε το τι γίνεται στην πράξη. Και δεν είναι σωστό να εξηγούμε στην συμφωνία το τι σημαίνει διαχωρισμός των εξουσιών, δίκη πρόσβαση στην δικαιοσύνη, ενώ ταυτόχρονα εντός της χώρας έχουμε δίκες πολιτικών αντιπάλων με διάφορες κατηγορίες, αλλά κυρίως για την πολιτική τους δραστηριότητα, που φοβούνται για την πρόσβασή τους στην δικαιοσύνη, που στερούνται το δικαίωμα σε δικαίη δίκη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά να τονιστούν στους Αρμενίους εταίρους σας ότι αυτά είναι βασικά σημεία της σύνδεσης με την Ευρώπη. Και δεν είναι σωστό να μιλάμε για χρηστή διοίκηση και μετά να μην παίρνουμε στα σοβαρά τις πραγματικές κατηγορίες διαφθοράς. Δεν είναι σωστό να μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη και να μην υπάρχει βασική προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Και βλέπουμε το πώς η μη διασφάλισή τους, ξεκινώντας με τα εργασιακά δικαιώματα και πηγαίνοντας στην ισότιμη εκπαίδευση, ακριβώς ε, εδρεώνουν ε, την εξουσία και αναπαράγονται συνεχώς ε, και στις εκλογές. Αυτά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχετε κατά νου, αλλά και στο τι συμβαίνει επί τόπου. Και βεβαίως ε, να γίνουν οι αλλαγές για τις οποίες δεσμεύεται ε, η κυβέρνηση, γιατί δεν σημαίνει αυτό. Και ευχαρίστως να απαντήσω και σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, εάν έχετε. Αυτά. Thank you, Ms. Ευχαριστούμε κυρία Μιναζιάν και τώρα περνάμε στην κυρία Λέβα η οποία θα μας μιλήσει για το Αζερβαϊτζάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 2006 και οι τρεις ε, δημοκρατίες του Νοτιού Καυκάσου ε, υπέγραψαν σχέδια δράσης ε, και είχαν και οι τρεις ε, μία ρήτρα πηγή έπνευσης για την ευρωπαϊκή τους φιλοδοξία. Στο Αζερβαϊτζάν είχαμε και μια εκστρατεία από πλευρά τη κοινωνία των πολιτών όταν ανακάλυψαν ότι για κάποιο λόγο δεν υπήρχε συγκεκριμένη ρήτρα. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτή την ε, δεκαετία ε, και μάλιστα το Αζερβαϊτζάν ε, δεν είχε καθόλου μείωση στο δημοκρατικό του έλλειμμα και απέκλεινε και από αυτή την ε, ενθουσιώδη δήλωση και την εφαρμογή της στη συνέχεια. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο διαρθρωτικούς παράγοντες. Ο ένας ε, μάλιστα ήταν και ε, ζηματική σημασία. Σίγουρα η περίπλοκη γεωπολιτική κατάσταση, η παρουσία εναλλακτική δύναμης της Ρωσίας και οι χώρες οι οποίες είναι απομονωμένες για την κατάσταση της Ρωσίας διότι δεν υπάρχει ένα αντίβαρο, ε, δεν υπάρχει μια ισχυρή δύναμη από τη Δύση ε, και από οποιονδήποτε άλλο εταίρο και επομένως ε, οι πιέσεις της Ρωσίας εξακολουθούν να είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγων ο οποίος καθορίζει και τη συμπεριφορά και την τακτική της χώρας. Η πίεση αυτή στο Αζερβαϊτζάν εφαρμόζεται, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, μέσω σειράξεων και από την αρχή της δεκαετίας του 90 ε, και εξακολουθεί να είναι και συνήθως ε, πραγματικότητα. Το Αζερβαϊτζάν τιμωρείται για τις ανεξάρτητες φιλοδυτικές πολιτικές ε, που επιδεικνύει από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέσω αυτής της πίεσης. Το άλλο διαρθρωτικό θέμα είναι εσωτερικό και εσωτερικό είναι η πολιτική οικονομία του πετρελαίου. Όλοι γνωρίζουμε ε, το παράδοξο της αυθονίας, ε, όλοι γνωρίζουμε τι παθαίνουν οι χώρες όταν ε, ξεκινούν εκτεταμένη εμπορική εκμετάλλευση του πετρελαίου ε, αμέσως μετά από την απομάκρυνση από την απεικιοποίηση όταν είναι ακόμα ισχνές οι πολιτικές ε, δυνάμεις και ε, το κράτος δικαίου και φυσικά τι γίνεται με όλα αυτά τα ενεργειακά συμφέροντα. Στην περίπτωση του Αζερβαϊτζάν μετά από το 2006 διότι τότε ξεκίνησε η μεγάλη εισρωή εισοδημάτων αυτό φυσικά ε, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης και πολύ συχνά υπάρχει και αυτό το οποίο αποκαλείται εθνικής των πόρων. Ε, δεν επιτρέπει δηλαδή την καλύτερη ολοκλήρωση. Εδώ αναφερόμαστε βεβαίω στο κατεστημένο και όχι στην κοινωνία. Και έρχομαι στο τρίτο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά τον τρόπο ε, συνεργασίας και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερβαϊτζάν. Φοβάμαι ότι η λεγόμενη διαφοροποίηση δεν έλαβε υπόψη της ε, αυτά τα διαρθρωτικά στοιχεία της οικονομίας δεν ε, κατάφερε να αντιμετωπίσει τα μεμονωμένα εμπόδια που αντιμετωπίζει κάθε χώρα για μεταρρύθμιση και σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, υπήρχε προφανώς από τη δεκαετία του 90 το θέμα της ανάπτυξης ασυμμετρίας ε, μεταξύ της κοινωνίας και του κράτους. Το κράτος ενισχύθηκε πάρα πολύ από την ε, πάρα πολύ μεγάλη εισρωή επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα ε, που ήταν και υποκρατικό έλεγχο και ε, ταυτόχρονα η κοινωνία ε, υποχρηματοδοτήθηκε και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αν δείτε και τους δυναμικούς συσχετισμούς θα δείτε ότι η κοινωνία των πολιτών του Αζερβαϊτζάν βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο, 10 φορές χαμηλότερο και από τη Γεωργία, πολύ χαμηλότερο και από την Αρμενία ίσως, της στήριξης για την κοινωνία των πολιτών. Ε, αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία των πολιτών έγινε πάρα πολύ ευάλωτη μέχρι το τέλος της δεκαετίας και επομένως το 2014 ε, είχαμε αυτή την τόσο δραματική ε, εξέλιξη και πίεση προς την κοινωνία των πολιτών όταν οι βασικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για ανθρωπιστικά δικαιώματα αλλά και άλλες έκλεισαν. Και ε, αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι πώς ε, το ενεργειακό θεματολόγιο, γνωρίζετε ότι το 2006 υπεγράφει το μνημόνιο για την ενέργεια και ουσιαστικά ε, το όλο θεματολόγιο της ενέργειας επηρέασε και το θεματολόγιο των ε, μεταρρυθμίσεων στο Αζερβαϊτζάν το Αζερβαϊτζάν, ή μάλλον το κατεστημένο το Αζερβαϊτζάν, ε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ε, το γόητρο μπορεί να βασίζεται μόνο στην οικονομική απόδοση. Και αν κάποιος αποκτήσει ε, πολύ καλό ενεργητικό στα θέματα της ενέργειας και στην ασφάλεια εφοδιασμού, αυτό επαρκεί για να γίνει αποδεκτός, να αναγνωρίζεται και να θεωρείται ισότιμος εταίρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν ε, ε, αναφερόμαστε στο Ζερποϊτζάν το θέμα της προσαρμοστικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εδώ η προσαρμοστικότητα εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι χώρες στην ε, γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι αυτό έλειπε πάντα στη σχέση μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και η βασική προσέγγιση. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο απουσιάζει και είναι αυτή η προσέγγιση. Υποστηρίζουμε απόλυτα τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έλεγα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πολύ έγκαιρα ε, και πολύ εύστοχα αντιδρούσε στα όσα συνέβαιναν ε, στην περιοχή αλλά και στην ίδια τη χώρα, αλλά δυστυχώς ε, δεν το ακολούθησαν άλλες δράσεις και δεν υπήρξαν συνέπειες για τη χώρα. Για την κοινωνία μας λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε διάκριση μεταξύ κατεστημένου και κοινωνίας, ιδιαίτερα σε μια χώρα που είναι πλούσια λόγω πετρελαίου, η ελίτ υπάρχει ε, εις βάρος του εισοδήματος από το πετρέλαιο. Δεν ε, υπάρχουν εισοδήματα από τη φορολογία λοιπόν, υπάρχουν εισοδήματα από το πετρέλαιο. Και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Ε, περιμένουμε λοιπόν μια καλύτερη προσέγγιση παρά το γεγονός ότι η νέα ε, παγκόσμια στρατηγική η προσέγγιση της νέας παγκόσμιας στρατηγικής ε, αναφέρεται σε ρεαλισμό, σε πραγματισμό και πιστεύουμε ότι αυτός ο ρεαλισμός δεν σημαίνει ότι θα παραμελήσουμε πλήρως τα θέματα τα οποία ε, οδήγησαν στα πιο ισχυρά και μοναδικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αυτή την ήπια δύναμη δηλαδή. Επίσης, θα θέλαμε να σας ε, ε, προειδοποιήσουμε γιατί μπορεί να υπάρξει μίμηση. Ε, το θέμα της διακυβέρνησης και της τομεακής συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει τελικά και σε μεγαλύτερη χειραγώγηση της όλης διαδικασίας της δημιουργίας θεσμών. Γιατί οι ηγέτες μας έμαθαν ε, πώς να χρησιμοποιούν τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις προς όφελός τους. Διότι ενώ ο επισήμως λοιπόν μπορεί να θεωρείται ε, μεταρρύθμιση, αποκέντρωση, ε, απορρύθμιση ή κάποιος αντίστοιχος όρος. Στην πραγματικότητα δημιουργεί όλο ένα και πιο κεντρική ε, συσσόρευση δυνάμεων. Και φυσικά αυτό θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στις πιθανές συμφωνίες οι οποίες είναι υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Το Αζερβαϊτζάν χαρακτηρίζεται όπως γνωρίζετε, από το γεγονός ότι έχει το μεγαλύτερο αριθμό πολιτικών κρατουμένων. Εάν δεν είναι λοιπόν η Ευρώπη, αν δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρουμε σε ποιον να βασιστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως του κ. Μανιέτοφ, ε, είναι ακόμα στη φυλακή. Ε, δυστυχώς υπάρχουν και κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις. Ε, ε συλλαμβάνονται δημοσιογράφοι όπως ο κύριος Αουσέινοφ. Ε, είχαμε το θάνατο κάποιου στη φυλακή του Γκαλαντάρ, ο οποίος ήταν μπλόγκερ και δημοσιογράφος. Πέθανε στη φυλακή και υπάρχουν και ε, δολοφονίες εξοδικαστικές. Εφτά άτομα δολοφονήθηκαν σε μια υπόθεση προδοσίας ε, και ε, ε, έγινε και μια ταφή κρυφή από στρατιωτικούς. Επίσης, θα θέλαμε να σας προειδοποιήσουμε για το καθεστώς, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσει να καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία δεν θα έχει καμία λογοδοσία και καμία, ε, ε, κανένας όρος. Δεν θα υπάρχει καμία ευθύνη για παραβίαση πολιτικών όρων. Θα ήθελα λοιπόν, δεν ξέρω πόσα λεπτά έχω στη διάθεσή μου ακόμα, αλλά πέντε μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι Προφανώς ε, και η ενέργεια, η ασφάλεια και το εμπόριο θα είναι οι τομείς ε, στους οποίους ε, θα συμφωνήσουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Αζερβαϊτζάν. Αλλά όπως σας είπα, η ασφάλεια εφοδιασμού είναι ένας από τους βασικούς διαρθρωτικούς παράγοντες που δυστυχώς δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα για την δημιουργία δημοκρατικού πολιτεύματος. Θα πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε αυτά υπόψη και θα πρέπει ε, να ε, ε, περιληφθούν στη νέα συμφωνία με κάποιο τρόπο. Τώρα, για τις συστάσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πετήσετε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατομένων και την βελτίωση των συνθήκων στη χώρα ε, ελευθερία ε, ε, της έκφρασης και φυσικά και συνθήκες κράτησης πολιτικών κρατουμένων και να πείτε ότι αυτή είναι ικανή και συνθήκη για να δημιουργηθεί μια στρατηγική συνεργασία επίσης όρης. Διότι από ό,τι κατάλαβα αυτό προσπαθεί να επιτύχει η πλευρά του Αζερβαϊτζάν. Ισότιμη σχέση. Ισότιμη σχέση όμως δεν υπάρχει χωρίς να υπάρξει δέσμευση για διεθνείς υποχρεώσεις ε, και καθολικά ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης, θα πρέπει να ζητήσουμε ε, και κατάργηση του συστήματος καταχώρησης ενισχύσεων και δωρεών για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, καλύτερη νομοθεσία, να ζητήσει αμνηστία για όλες τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, να ε, αποδεσμεύσει τους λογαριασμούς τους, ε, να σταματήσουν οι απαγορεύσεις ταξιδίων και επίσης να διασφαλίσουν ότι θα συμμετέχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο διάλογο με το Αζερβαϊτζάν και επίσης ε, να αποκλείεται και ε, κάποιες ε, συμπεριφορές συγκεκριμένες. Επίσης, η προσχώρηση του, ε, του Αζερβαϊτζάν στον ΠΟΕ είναι μία από τις προτεραιότητες. Και επίσης, χρειαζόμαστε και πιο συγκεκριμένες διατάξεις, κίνδυνοι ε, για τομεακή συνεργασία, ε, οι παρούσε τάσει δεν θα έχουν πολύ σημαντικέ συνέπειες, Επομένω, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εγγυηθούμε διαφάνεια όλων των δράσεων οι οποίε θα προκύψουν από τη συνθήκη, θα πρέπει να πιέσετε για τομεακές ε, πολιτικές και σύγκληση σε θέματα νομοθεσία. και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίσει και τι εσωτερικές συνέπειε του θέματο τη ασφάλεια εφοδιασμού για τον προμηθευτή ε, στη χώρα και να δούμε και τι γίνεται στο θέμα της ασφάλειας ε, ε, εφοδιασμού στη χώρα. Να χρησιμοποιηθεί επίσης η εμπορική συνεργασία για να δώσουμε όθηση για μεταρρυθμίσεις και διαφοροποίηση της οικονομίας και αποκέντρωση και απελευθέρωση. Και φυσικά ένα από τα θέματα που αποτελεί πρόβλημα είναι ότι όταν υπάρχουν περιορισμένοι διάβλοι επιρροής ε, στον πολιτικό τομέα, θα πρέπει να προσπαθήσετε να αυξήσετε τη στήριξη για την παιδεία, τις πανεπιστημιακές και τις ε, επιστημονικές ανταλλαγές, ε, να συμμετέχουν σε πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα και μέσω ε, κατάλληλων δράσεων δημιουργίας δυνατοτήτων και εκστρατιών ενημέρωσης. Εδώ θα σταματήσω και θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας αν υπάρχουν. Thank you, Ευχαριστούμε κυρία Αλιέβα για την ενημέρωση σχετικά με το Αζερβαϊτζάν. Στο μεταξύ ο κύριος Δερκ Σιούμπελ έχει φτάσει. Ε, συνάδελφοι, θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Σιούμπελ και στη συνέχεια έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για ερωταποκρίσεις και συζήτηση. Το γνωρίζετε τον κύριο Σιούμπελ φυσικά, είναι ε, υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις των κλαδικών μερών και των δύο συμφωνιών. Έχετε το λόγο κύριε Σιούμπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα, συνάδελφοι. Φίλοι της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, λυπάμαι που άργησα. Είναι μια ε, μέρα πολύ γεμάτη σήμερα. Μόλις τώρα τα κατάφερα να έρθω και έχασα μέρος των παρουσιάσεων. Έφτασα μόλις στο τέλος. Θα ήθελα όμως να σας δώσω τη δική μας προοπτική από πλευρά της ΕΙΕΘ που βρισκόμαστε για τις δύο χώρες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις νέες συμφωνίες. Ξεκινώντας με την Αρμενία. Όπως γνωρίζετε, ανακεφαλαιώνοντας λίγο ιστορικά, ήταν πρώτη μέρα στο γραφείο ε, με την ιδιότητά μου στις 3 Σεπτεμβρίου του 2013, όπου η Αρμενία αποφάσισε να αποσυρθεί από την συμφωνία που είχε ε, τύχει διαπραγμάτευσης και έλεξε να ενταχθεί στην Ευρωασιατική Οικονομική Συνεργασία αλλά είπαμε ότι θα, θέλαμε να συνεχίσουμε μια στενή σχέση με την... Ε, είπε ότι θα, ήθελα να συνεχίσει στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χωρίς ε, συμφωνία σύνδεσης. Πήρε χρόνο να σκεφτούμε τι ε, θα ήταν δυνατόν πολιτικός και τεχνικός με αυτή τη μορφή. Μετά από 18 μήνες περίπου περιμέναμε τις απόψεις της Αρμενίας. Επ' αυτού η Αρμενία έπρεπε να ε, δει ποιες ήταν οι δεσμεύσει ε, με την ένταξή της στην Ευρασιατική Οικονομική Συνεργασία. Και εν τέλει το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ε, μια νέα εντολή διαπραγμάτευσης για αυτή την συμφωνία και ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2015 οι διαπραγματεύσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν ε, σύντομα, ε, δεδομένου ότι είναι νέα συμφωνία, τον Φεβρουάριο του 2017. Ε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν θέματα τα οποία είχαν ήδη συζητηθεί και λάβαμε υπόψη ε, τα θέματα των προηγούμενων ε, διαπραγματεύσεων και των τομεακών μερών και χαρήκαμε που η Αρμενία συμφώνησε με ε, πολλά από τα μέρη της νομικής προσέγγισης και ήταν έτοιμη να συμφωνήσει και να υλοποιήσει μέσα από αυτή τη συμφωνία αρκετά από αυτά τα θέματα για κάποιους τομείς δώσαμε μεγαλύτερη προθεσμία για την υλοποίηση, αλλά συνολικά νομίζω είναι μια καλή συμφωνία, φιλόδοξη. Βέβαια, ε, το DCFTA, το εμπορικό κομμάτι, είναι λιγότερο φιλόδοξο τώρα, λόγω του γεγονότος ότι φυσικά ε, υπάρχει ευρωασιατική συνεργασία που έχει αρκετές απαιτήσεις που δεν μπορούν να ε, ταιριάσουν με τις απαιτήσεις του DCFTA. Αυτό που κάνουμε ε, τώρα με αυτή τη νέα συμφωνία, η συμφωνία λέγεται συνολική και ενισχυμένη ε, συμφωνία εταιρικής σχέσης, συνολική και ενισχυμένη, η ΣΕΠΑ είναι το ακρονίμιο, ξεκίνησε τον Μάρτιο και τώρα ετοιμάζονται οι η φάση της, ε, των υπογραφών. Ε, γίνεται η επαλήθευση του κειμένου από τους ε, νομικούς γλωσσολόγους μας, μετάφραση σε όλες τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα αρμανικά και όλες οι άλλες διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσουν και οι δύο πλευρές έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Εάν ολοκληρωθούν όλα αυτά τα βήματα, η ΣΕΠΑ μπορεί να υπογραφεί ε, στο περιθώριο της, της Συνόδου Κορυφής τον Νοέμβριο της, ε, των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Ε, είναι δυνατόν να υπάρχουν βαθιές και ευρείες σχέσεις με ε, τις χώρες που ανήκουν και στη βρασιατική συνεργασία. Ένα από τα κλειδιά στην επιτυχία της διαπραγμάτευσης είναι ότι δώσαμε ε, προσοχή στις άλλες διεθνείς ε, δεσμεύσεις της Αρμενίας. Η ΣΕΠΑ, σε αντίθεση με την Συμφωνία Σύνδεσης που υπήρχε προηγουμένως, δεν περιέχει την ευρεία ζώνη ε, εμπορίου. Ε, δεν... Αυτό θα ήταν διαφορετικό ε, αν ήταν στα πλαίσια του DCFTA. Νομίζω τα περισσότερα τα έχω αναφέρει. Πιστεύουμε ότι θα, ολοκληρω ότι αυτή η συμφωνία δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον εμπορίου και επενδύσεων, παρόλο που δεν περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τις επενδύσεις όταν υπογραφεί. Αυτά σχετικά με την Αρμενία. Τώρα, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, βεβαίως δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ όσο προχωρήσαμε στο, στην, συμφωνία με την Αρμενία. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης το 2011 2012 Ωστόσο, συνειδητοποίησαμε ότι το Αζερβαϊτζάν δεν ενδιαφερόταν ε, για μια τόσο στενή σύνδεση όπως άλλες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το Αζερβαϊτζάν ήθελε ε, μια σχέση ίσων εταίρων με βάση ε, το αμοιβαίων όφελος. Αυτό ληφθεί υπόψη στη, στη Σύνοδο Κορυφής της Ρήγας το 2015 και ο Υπουργός Εξωτερικών είχε παρευρεθεί με τον ε, Επίτροπο ε, Χάν και ε, και εξέφρασε το ενδιαφέρον να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις επί ενός νέου κειμένου μιας συμφωνίας σύνδεσης που θα διεύρυνε το πεδίο εφαρμογή των σχέσεών μας δεδομένου ότι η PCA είναι 20 χρόνων τώρα, είναι παροχημένη γι' αυτό χρειάζεται μια καινούρια βάση και λαμβάνουμε υπόψη επίσης και την αναθεώρηση της, επιτρο... της ε, πολιτικής γειτονίας και των οικονομικών προκλήσεων που έχουν προκύψει από τότε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλησε εις βάθος το κείμενο και είχε και μια αποστολή στο Μπακού το 2015 για να ορίσει το πεδίο εφαρμογή μιας μελλοντική συμφωνίας ε, και τα κατακόλουθα. Πρώτα απ' όλα το επίπεδο φιλοδοξίας δεν πρέπει να κάνω κάτω από ε, την ε, σημερινή συμφωνία σύνδεσης. Πρέπει να είναι δεσμευτικές, νομικά δεσμευτικές. Η νέα συμφωνία θα πρέπει να αντικαταστήσει την τερέχουσα συμφωνία τερικής σχέσης και σύνδεσης και ήταν ενδιαφέρον διότι σύμφωνα με τις ε, ε, γνώσεις που έχουμε, ήταν η πρώτη φορά που τρίτη χώρα παρουσιάζει σχέδιο συμφωνίας στην ΕΕ. Άρα αυτό απέτησε κάποια ευελεξία από δική μας πλευρά για το πώς θα κινούμασταν, πώς θα το χειριζόμασταν αυτό το σχέδιο, γραφειοκρατικά μιλώντας. Βρήκαμε μια καλή λύση όμως. Πήραμε μέρη ε, της πρότασης του Αζερβαϊτζάν όταν ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη που ε, πήραμε στις 14 Νοεμβρίου περασμένου χρόνου, όπου το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε αυτή την εντολή και έχει ε, διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή των σχέσεων. Λάβαμε υπόψη την αναθεώρηση της ευρωπαϊκή πολιτικής γειτονία και αυτά που είπα προηγουμένω. Οι διαπραγματεύσει ε, ξεκίνησαν πριν, ε, στις 7 Φεβρουαρίου του 2017 και στο περιθώριο της μιας επίσκεψης του Προέδρου Αλιεύ στις Βρυξέλλες. Η έναξη των διαπραγματεύσεων παρέχουν ένα παράθυρο ευκαιρίαση για την επικαιροποίηση της νομικής βάσης και της κατάστασης πραγμάτων των σχέσεων μας. Θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τους τομείς συνεργασίας μας. Αν δείτε υπάρχουν ε, τομείς που δεν καλύπτονταν επαρκώς στο παρελθόν, στην προηγούμενη συμφωνία. Ε, βεβαίως παρέχεται και μια ευκαιρία διεύρυνση τη συνεργασία ε, αυτή τη στιγμή που το Αζερβαϊτζάν προσπαθεί να διαφοροποιήσει την οικονομία ε, πέραν από τον ενεργειακό τομέα που είναι η πρώτη προτεραιότητα βέβαια στην οικονομία του Αζερβαϊτζάν έχει εκφράσει ενδιαφέρον να συνεργαστεί και σε άλλους τομείς μεταφορές για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα το Αζερβαϊτζάν βρίσκεται στο σταυροδρόμιο ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Τουρισμός, ένας άλλος τομέας, ε, καταπολέμησης τρομοκρατίας, ψηφιακή οικονομία, που τώρα στα πλαίσια της εσωνικής προεδρίας αναφέρθηκε ε, επανειλημμένος. Επίσης, και για να σχολιάσω στα σχόλια της κυρίας Αλίεβα, παρέχει μια ευκαιρία επικαιροποίησης της δέσμευσης ε, του Αζερβαϊζάν για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τουλάχιστον για αυτά που προέρχονται από την ιδιότητά του ως μέλος του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι σημαντικό. Το συζητήσαμε ήδη με τα κράτη-μέλη όταν διαπραγματευτήκαμε και συμφωνήσαμε ε, για αυτή την εντολή. Η συμφωνία θα καλύπτει βέβαια κλασικά ε, πολιτικά, νομιακά, εμπορικά μέρη οικονομικά μέρη θα έχει ένα τίτλο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διοίκηση που ε, το έχει χαιρετήσει το Ζερμπαϊζάν και οι διαπραγματεύσεις όπως ε, και άλλες διαπραγματεύσεις που έχουμε με τρία ε, χρόνια καλύπτονται από τρεις ομάδες εργασίας, μία για πολιτικά θέματα από τον επικεφαλής διαπραγματευτή τον Λουκ Ντεβινιέ τον Διευθυντή μου των Εξωτερικών Σχέσεων που έχει διαπραγματευτεί και για το θέμα της Αρμενίας, η δεύτερη ομάδα ε, για θέματα εμπορίου και, τρίτη ε, εβδομάδα, ε, και η τρίτη ομάδα επίσης. Μέχρι στιγμή έχουμε κάνει δύο γύρους διαπραγματεύσεων για το πολιτικό μέρος, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Θα ακολουθήσει και τρίτος γύρος πριν από το καλοκαίρι και υπάρχει δέσμευση και από τις δύο πλευρές να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις στο συντομότερο δυνατόν και στο πολιτικό μέρος να πούμε ότι έχουμε τους τίτλους για τον πολιτικό διάλογο, τον τίτλο των ανθρωπινών δικαιωμάτων, ε, δικαιοσύνη, ελευθερία και ε, ασφάλεια. Έχουμε κάνει καλή πρόοδο, πρέπει να σας πω, και ε, στο θέμα των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Δεν απέχουμε πολύ από μια γενική συμφωνία. Στην ομάδα εργασίας για θέματα εμπορίου είχαμε ένα γύρο τον Ιούνιο και το έργο συνεχίζεται ε, με βίντεο ε, συσκέψεις, τηλεσυσκέψεις. Ε, διαπραγματεύσεις έγιναν για τα θέματα διαφάνειας, SPS, τελωνία, πνευματική ιδιοκτησία και θα υπάρχουν 12 διαφορετικά κεφάλαια στο, στο θέμα του εμπορίου. Βέβαια, η μη ένταξη στον ΠΟΕ δεν βοηθάει. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε εάν ήταν μέλος του ΠΟΕ. Ελπίζουμε ότι θα εντείνουμε το έργο μας και θα συμβάλλουμε επίσης και ε, να βοηθήσουμε το Αζερβαϊτζάν να ενταχθεί ε, στην συνεργασία την κλαδική. Ξεκίνησαμε δύο γύρους, ανοίξαμε μια κεφάλαια, κλείσαμε ήδη τρία και πάλι σε αυτό το μέρος θα έχουμε ένα κεφάλαιο για την κοινωνία των πολιτών. Δεν έχει ακόμη ανοίξει, θα ανοίξει όμως. Και η νέα συμφωνία, αφού ε, κλείσουν οι διαπραγματεύσεις, θα αποτελεί μια καλή βάση για περαιτέρω εντατικοποίηση των σχέσεων με το Αζερβαϊτζάν, τηρουμένων όλων των θεμάτων που έχουν εγερθεί από την ΕΛΕ Θα κλείσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Right, thank you, Mr. Σας ευχαριστώ, κύριε Ακούσαμε τρεις ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Και νομίζω ότι έχουμε τώρα την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις ε, και συζήτηση. 45 λεπτών θα έλεγα. Λοιπόν, έχουμε συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το Αζερβαϊτζάν και άλλους για την Αρμενία. Δεν έχει νόημα να τα χωρίσουμε. Οπότε θα δώσω τον λόγο στους συναδέλφους που ζήτησαν να μιλήσουν. Τρία λεπτά ο καθένας. Ωραία. Ωραία. Σόφκο από το ΕΛΚ. Λοιπόν, πρώτη, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για το Ζερβαϊτζάν, μια που είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Η νέα συνολική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αζερβαϊτζάν θα πρέπει να αποτελέσει ένα μέσο συνεργασία για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντο και κοινών στόχων, όπως η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση πηγών ενέργεια. Επίση, η συνολική συμφωνία αναπτύσσεται για αυτά τα ζητήματα και δεν θα πρέπει όμως να παραμερίζει τις βασικές αξίες των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης. Τούτου λεχθέντος αναγνωρίζω την συμφωνία των αρχών, τη σημασία με συγχωρείτε των αρχών δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας παρά το ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και δημοσιογράφων ε, και η νομοθεσία περί κοινωνίας των πολιτών έχει αλλάξει. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει όπως φαίνεται και από την πρόσφατη φυλάκιση του Αφγάν Μουφτάρη, του δημοσιογράφου και άλλων, για να γίνει το Αζερβαϊτζάν αξιόπιστος εταίρος της Ένωσης. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας όσον αφορά τις νέες εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών. Όλοι γνωρίζουμε πως η σύγκρουση του Ναγκόρν Καραμπάχ θα πρέπει να επιληθεί χωρίς στρατιωτικά μέσα. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια πολιτική λύση στην σύγκρουση αυτή. Στηρίζω τις ε, προτάσεις ε, της ομάδας του Μίνσκ του ΑΣΕ. Και πρέπει να πω ότι προσφάτως πήγα σε μια αντιπροσωπεία της ε, ΑΦΕΤ σε Αρμενία και Γεωργία και κατά την ταπεινή μου γνώμη θεωρώ ότι χωρίς διάλογο δεν μπορούν να βοηθηθούν αυτές οι χώρες για να, να επιτύχουν ειρήνη και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα ηθικό ανάστημα για να βοηθήσει. Σας ευχαριστώ και απευθύνω έκκληση στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να βοηθήσει τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών. Χοβάλα. Τώρα θα ακούσουμε κάποιον από τους σοσιαλδημοκράτες. Κανείς. Μάλιστα. ECR, Charles Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω η ομάδα μου στηρίζει την συμφωνία σύνδεσης με το Αζερβαϊτζάν και προφανώς το παρελθόν είχαμε ασκήσει κριτική για την έλλειψη δημοκρατίας, και γενικά τον τρόπο διοίκησης ε, του Μπακού και βέβαια υπάρχει και το θέμα με την Αρμενία. Εγώ Βεβαίω λυπήθηκα, αλλά αντιλαμβάνομαι γιατί η Αρμενία δεδομένης και της κατάστασης με την Ρωσία δεν μπορούσε να υπογράψει την συμφωνία εκείνη τη στιγμή και θεώρησε ότι καλό ήταν να πάει ε, προς την κατεύθυνση της ε, ευρασιατικής οικονομικής κοινότητας υπό την ομπρέλα της Ρωσίας. Έκτοτε όμως δεν ε, ξέρω αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στην Ευρασιατική Ένωση. Φαίνεται ότι είναι σε ένα εμβριακό στάδιο και μάλλον περισσότερο βρίσκεται ε, στο επίπεδο των συμβολισμών. Αλλά τέλος πάντων προφανώς αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Είναι θέμα των Αρμενίων και της Μόσχας. Αλλά θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο θέμα το μεγάλο το οποίο όλοι αποφεύγουμε. Και βεβαίω ίσως δεν μπορούσαν οι ειδικοί από τις δύο χώρες να το θίξουν. Ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να μιλήσει ε, στην κλιμάκωση που είχαν πρόσφατα στη γραμμή αντιπαράταξης με τον τραγικό χαμό δύο αμάχων νομίζω. Και στο παρελθόν είχαμε ε, Αρμένιους που σκότωσαν ελεύθεροι σκοπευτές κτλ. Πώς μπορούμε να αποκλιμακώσουμε την σύγκρουση, πώς μπορεί η διαδικασία του Μίνσκ του ΟΑΣΕ να βοηθήσει. Και το ερώτημα που κάνω βεβαίω είναι κατά πόσον θα πρέπει να βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία του Μίνσκ αντί για την γαλλική κυβέρνηση και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστείλει μια αποστολή παρακολούθησης ε, στα σύνορα αντί για τον ΟΑΣΕ. Υπάρχει κάποιος ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Το έχουμε συζητήσει πριν από μία δεκαετία, αλλά δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Νομίζω ότι υπάρχει τώρα μια ευκαιρία για την κυρία Μογκερίνη να δραστηριοποιηθεί. Και προφανώς ε, βεβαίω χρειάζεται και συνεργασία του Παρισίου και των Γάλλων, γιατί αυτοί έχουν εμπλακεί στην διαδικασία, αλλά έχουν εντύπωση ότι το Μίνσκ δεν έχει αποτελέσματα η διαδικασία αυτή. Και υπάρχει ακριβώς ο κίνδυνος ε, στην γραμμή αντιπαράταξης ε, που υπήρχε πριν από μία δεκαετία. Σας ευχαριστώ. Από την Άλντε έχουμε τέσσερις συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Ξεκινάμε με την κυρία Νικολάη που είναι η συγγήτρια για το Αζερβαϊτζάν. Σας ευχαριστώ. Εγώ... Εγώ καλωσορίζω και τις δύο συμφωνίες αυτές ε, και με την Αρμενία και με το Αζερβαϊτζάν είναι μια καλή ευκαιρία για να είμαστε παρόντες και οπωσδήποτε έχουμε κάποιες διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Η μία χώρα είναι πιο κοντά στη Ρωσία, η άλλη θέλει να απομακρυνθεί από τη Ρωσία. Αλλά ελπίζω αυτό να μην αποτελέσει εμπόδιο για τις εξελίξεις στην περιοχή. Για εμένα το βασικό πρόβλημα είναι η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή και λυπούμε ιδιαιτέρως ε, για το περιστατικό της 4ης Ιουλίου όταν δύο ε, γυναίκες ε, αζέρισες σκοτώθηκαν από τον αρμενικό στρατό. Πρόκειται για μια κλιμάκωση και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και από τα δύο μέρη να σταματήσουν την βία στα σύνορα γιατί το συμβάν της 4ης Ιουλίου δεν ήταν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ήταν στην επικράτεια του Ζερβαϊτζάν. Κάποιο είδου επίθεση δηλαδή θα έλεγα, μια επιθετική ενέργεια. Μας ανησυχεί λοιπόν το τι συμβαίνει στην περιοχή, γνωρίζουμε το τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ζητάμε αυτά, πάντα ζητάμε βελτίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό θα αποτελέσει μέρος της πολιτικής μας προσέγγισης και θεωρώ ότι το συντομότερο ε, δυνατόν θα πρέπει να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία και όσο συντομότερο τόσο το καλύτερο γιατί έτσι θα μπορέσουμε να διαδώσουμε τις αξίες μας στην περιοχή καλύτερο αυτό από το να ασκούμε συνεχώς κριτική και καλό είναι να υπάρχει ε, και η συνεργασία. Και ελπίζω μετά να είναι πιο παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί για εμένα έχει αποτύχει ε, η διαδικασία του Μίνσκ. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Μιλάμε και χρόνια ε, και δεν έχουμε κανένα από το αποτέλεσμα. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελέσει μέρος ενός συμφώνου σταθερότητας στην περιοχή, νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό για να έχουμε κάποια σταθερότητα στην περιοχή, σεβόμενοι τα δικαιώματα αυτοδιάθεσης ε, του Αζερβαϊτζάν. Καλωσορίζω λοιπόν αυτήν την ε, συζήτηση και ελπίζω αν ε, συνεργαστούμε να έχουμε κάποια βελτίωση στην ε, καθημερινή ζωή των πολιτών ε, του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Σας ευχαριστώ. Με τον κατάλογο που βλέπω έχουμε πέντε ομιλητές ακόμα. Γκάλ, Κιούρε, και Νάτ. Και τον κύριο Μπούχνερ. Μου ξέφυγε κάποιος. Λοιπόν, τελειώνει εδώ ο κατάλογος. Λοιπόν, κύριος Γκάλερ τώρα. Σας ευχαριστώ για μένα είναι πολύ ε, επίκαιρη η στιγμή γιατί την Πέμπτη πηγαίνω στην Αρμενία σε ένα συνέδριο. Θα επικεντρωθώ λοιπόν στην Αρμενία και θα προσπαθήσω, θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς δηλαδή, πώς ακριβώς ε, σκοπεύει η χώρα σας να εφαρμόσει ε, τα όσα έχουν υπογραφεί αν σκεφτούμε τα όσα έγιναν. Είχαμε τη συμφωνία, άλλοι την είχαν υπογράψει, άλλοι όχι. Να το συγκρίνουμε λοιπόν το ερώτημά με το εξή. Οι Αρμένοι τότε, ε, δεν ξέρω, ίσως σας είπε ξεκάθαρο ο κύριος Πούτιν ότι αν υπογράψετε ε, δεν θα έχετε την ε, στήριξή μου την στρατιωτική για το Αζερβαϊτζάν. Οπότε το σκεφτήκατε κι εσείς και το είδατε κάπως λιγότερο φιλόδοξα. Για να ρωτιέμαι, μήπως. Εντάξει, όχι ίσως το εμπορικό, αλλά το πολιτικό κομμάτι να το δείτε κάπως πιο μακροπρόθεσμα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή για την δημοκρατική εξέλιξη της χώρας. Είναι τελείως διαφορετική η εξέλιξη από το όσο σκεφτόμασταν το 2013. Τότε ήταν ο κύριος Γιάννου Κόβιτς. Ε, φαντάζομαι και αυτός θα ήθελε να επικεντρωθεί περισσότερο στην οικονομία. Ε, περισσότερο, γιατί η δημοκρατία και τα λοιπά, όλα ίσως να μην τα είχε σκεφτεί τόσο. Οπότε είναι και θέμα πολιτικής βούλησης ε, για να εφαρμόσουμε τα όσα υπογράφουμε. Εσείς πώς θα το εκτιμούσατε, μια χώρα όπως η Αρμενία όταν υπογράφει μια τέτοια συμφωνία μήπως ε, το συνδέει και με την ε, συνταγματική μεταρρύθμιση και με το να επιτύχει μια συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν θεωρείται ότι έτσι έχει ενισχυθεί τόσο πολύ ώστε να εμπλακεί περισσότερο με την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκάλεα. Γιούρεκ για το ECR για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μια ειρηνική λύση της ε, σύγκρουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά δυστυχώς οι προποθέσεις ε, για αυτή την ε, λύση είναι να διατηρηθεί η κατάπαυση πυρός και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μηχανισμός ο οποίος να μας επιτρέπει να παρακολουθούμε κατά πόσον τηρείται η Συμφωνία κατάπαυση Πυρός, παρά το γεγονό ότι η ομάδα του Μίνσκ έχει κάνει επανειλημμένες εκκλήσει για τη σύσταση ενό τέτοιου μηχανισμού. Ε, ανεξάρτητα από το τι ε, άποψη έχουμε για τις ε, θέσεις της ομάδος, η πρότασή τους είναι πάρα πολύ καλή για να αποφύγουμε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Ξέρουμε ήδη ότι τον περασμένο μήνα είχαμε ένα περιστατικό το οποίο η Ερμονία θεωρεί ότι ήταν προσχεδιασμένο διότι ε, έγινε σε κατοικημένη περιοχή. Επομένως, εάν θέλουμε να έχουμε μηχανισμούς που θα προλαμβάνουν τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να κάνουμε κάτι. Ε, μια συγκεκριμένη πρόταση, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, είναι να κάνει μια έκκληση η ύπατη εκπρόσωπος ε, στις δύο πλευρές ε, να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό τον οποίο προτείνει η ομάδα του Μίνσκ. Τώρα, όσον αφορά τις ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών και σύνδεσης με τις δύο χώρες, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτό ως όρο καλής θελήσεως, δηλαδή να δεχτούν την πρόταση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να αναλάβει πρωτοβουλία, είπατε εκπρόσωπο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάγγελ για τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι παράδοξο το γεγονός ότι συζητάμε νέες συμφωνίες με δύο χώρες, οι οποίες είναι όμορες χώρες και ταυτόχρονα πάρα πολύ διαφορετικές. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση και η εμπειρία ε, από τις απόπειρε προηγούμενων συμφωνιών με τις δύο χώρες μας έχει διδάξει ότι ίσως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την συγκεκριμένη γεωγραφική τους θέση, τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά που έχουν η κάθε χώρα και τη θέση τη δική μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι στη δική μας την περίπτωση, όταν αναφερόμαστε στα δικά μας τα συμφέροντα και το ενδιαφέρον για ειρήνη και σταθερότητα ε, στην ε, άμεση γειτονία μας, τότε σίγουρα το Αζερβαϊτζάν είναι μία από τις χώρες ε, που βρίσκεται πιεσμένη ανάμεσα στις δύο μεγάλες ε, όμορες χώρες που έχουν πολύ μεγάλα στρατηγικά συμφέροντα. Από τη μια έχει το Ιράν στο νότο και από την άλλη έχει τη Ρωσία ε, στα βόρεια. Η Αρμενία έχει λάβει τις αποφάσεις της και έχει μόνο ένα στενό φίλο και υποστηρικτή ε, θυμάμαι άλλωστε τη δήλωση του Προέδρου της Αρμενίας, ο οποίος είπε ότι η παρουσία των ρωσικών ε, στρατευμάτων ε, στην επικράτειά μας αποτελούν την πιο σημαντική εγγύηση ασφαλείας για μας. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι υποδιαπραγμάτευση δύο συμφωνίες σίγουρα αποτελεί ένα θετικό βήμα, σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε βελτίωση των συνολικών σχέσεων στην περιοχή και θα μπορούσε ίσως να βελτιώσει και την ε, ε, δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, και οι δύο παρατηρήσεις που έγιναν από τους ομιλητές για τα θέματα αυτά ήταν πολύ επίκαιρες και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά να πω και το εξή. Δεν βλέπω ενδεχόμενο σταθερή ε, σχέσης εάν δεν αντιμετωπιστεί το θέμα του Γκόρνο Καραμπάχ ε, με ε, μεγαλύτερη σοβαρότητα. Ε, ακούω τι λένε οι συνάδελφοι για τις προτάσεις της ομάδας του Μίνσκ πιστεύω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο και στην ίδια την ομάδα του Μίνσκ. Ε, ε, εμείς κάπως πριν από χρόνια Εγκαταλείψαμε την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ομάδα του Μίνσκ και τη δώσαμε στη Γαλλία. Ε, δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτά όλα οδηγούν σε πιο δραστήριο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την επίλυση του προβλήματος. Επίσης, ε, θα ήθελα να επισημάνω και το εξής. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η μόνη λύση ε, για αυτή τη μορφή τα προβλήματα είναι μέσω διεθνούς δικαίου. Και το διεθνές δίκαιο ε, σε αντίστοιχες περιπτώσεις αναγνωρίζει ε, μη χώρα ως χώρα κατοχής και ε, τη χώρα της οποίας τα εδάφη είναι υποκατοχή. Θα πρέπει λοιπόν να το πούμε και στις δύο πλευρές σαφέστατα και σε αυτή την περίπτωση και ίσως αυτές οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν και μία ευκαιρία για μας για να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και στις δύο πλευρές ότι χρειάζεται ε, μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για να μπορέσουν να έχουν σχέσεις καλής γειτονίας ε, και κατανόηση ο ένας προς τον άλλον. Η κρατική προπαγάνδα δεν έχει αποτελέσματα σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βάγκελ. Ο κύριος Μπούχνερ τώρα. Ευχαριστώ. Δύο σύντομες ερωτήσεις έχω εγώ. Η πρώτη είναι το Αζερβαϊτζάν δεν είναι μέλος ε, του ΠΟΕ. Πότε αναμένεται να γίνεται να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, και να γίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, για την Αρμενία. Μιλήσαμε βεβαίως για το ότι οι εμπορικές σχέσεις ε, περιορίζονται μέσω του ότι η χώρα εντάχθηκε στην Ευρασιατική Συνομοσπονδία. Ε, υπήρχαν και άλλες δυσκολίες με άλλες ε, χώρες, οπότε οποιασδήποτε λεπτομέρειες μπορούσατε να μας δώσετε, θα με ενδιαφέραν ιδιαίτερως. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι, ο κύριος Αουστρεβίτσιους. Ευχαριστώ Ευχαριστώ που οργανώσετε αυτή την ακρόαση και έχετε καλέσει και με κυβερνητικέ οργανώσει και από την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν και τον κύριο Σούμπερ. Μα δίνουν ε, πλήρε πληροφορίε για το πώ έχει κατάσταση. Έχουμε μία σύγκρουση η οποία έχει παγώσει, την οποία δεν δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά, αλλά από τη χώρα που βρίσκεται πιο βόρεια, που ήθελε να έχει και κάποιους μοχλούς πίεσης ε, έναντι όλων των χωρών του Νοτιού Καυκάσου. Και είναι πολύ εύκολο να διαχειρίζεσαι μια κατάσταση όταν έχεις κάποιες χώρες ε, υπόλογες ε, και έχεις και κάτι να τις πιέσεις. Τι εννοώ. Ούτε οι κατεχόμενοι, ούτε η χώρα που ε, είναι υπεύθυνοι για την κατοχή θα πρέπει ε, να ε, είναι ελεύθερες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να επικρίνουμε και τις δύο πλευρές. Η απόψή μας δεν έχει σχέση με το για ποια χώρα μιλάμε, την Αρμονία ή το Αζερβαϊτζάν η υποχρεωτική απαγωγή του κ. δεν είναι μήνυμα προς την ε, κυβέρνηση. Είπαμε στους Αζέρους μην το κάνετε, μην διαπράξετε αυτό το σφάλμα. Και το αυτό ισχύει και για την Αρμενία. Και όταν διαβάζω και τις εκθέσεις για την κατάσταση ε, στην περιοχή του Ορχανλή, ε, συγγνώμη, Λυπάμαι που είχαμε θύματα ε, από πλευρά Αζέρων, αλλά διαβάζω και την έκθεση της πλευράς των Αζέρων που λένε ότι ε, επιτέθηκαν σε ε, αρμενικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονταν εκεί κοντά. Δεν είναι λύση για να επιληθεί η σύραξη αυτή στην περιοχή. Τώρα, η ερώτησή μου προς εκπροσώπους των κυβερνητικών οργανώσεων. Πώς βλέπετε το διάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κάθε χώρα. Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόοδος στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αρμενία και το Τζερβοϊτζάν. Και η δεύτερη ερώτηση, πώς αξιολογείτε τις επαφές μεταξύ των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων μεταξύ των δύο χωρών. Δεν μιλούν οι θύνοντες στο βαθμό που θα έπρεπε. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, δηλαδή να έχουν ανθρώπινες επαφές ε, σε διαφορετικό επίπεδο. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Και ερώτησή μου προς τον ε, κύριο Σούμπελ. Έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις ε, με δύο χώρες, η μία είναι από την Ευρασιατική Ένωση και η άλλη είναι από την Κοινοπολιτεία των λεγόμενων ανεξαρτήτων χωρών. Ε, έχουμε ξεκινήσει λοιπόν αυτή τη συζήτηση εν μέρη ε, στην πραγματικότητα με την Ευρασιατική Ένωση. Δεν ξέρω τι γίνεται με το κεκτημένο της Ένωσης αυτής, ξέρω όμως τι γίνεται με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται με τη λογοδοσία. Ε, τι συνέπειες μπορούμε να δούμε στο μέλλον ε, για τι, πώς μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ και τέλος ο κύριος ε, Νάρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Αρμενία είναι περίεργη χώρα, σημαντική. Παρά το γεγονός ότι η δημογραφική αύξηση είναι θετική, ε, δημογραφικά όμως μειώνεται ο πληθυσμός της, διότι οι νέοι φεύγουν. Και οι νέοι, οι καταρτισμένοι νέοι φεύγουν από την Αρμενία γιατί δεν έχουν καμία εγγύηση για καλύτερη ζωή και δεν την έχουν γιατί η διαφθορά είναι ο ορισμός ε, και οι πολλαπλές ολιγορχίες οι οποίες μοιράζονται τον κάθε οικονομικό τομέα της χώρας είναι μία ακόμα από τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζει η χώρα. Όταν λοιπόν εγώ ακούω για πολιτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι πολύ διαρθρωτικές, όταν ε, η διαρθρωτική δομή της κοινωνίας είναι ανέγγιχτη, διότι ελέγχεται από τους ολιγάρχες ε, της κάθε περιοχής ε, ε, της χώρας, ε, ε, οι οποίες έχουν μοιραστεί την τούρτα με σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και δεν έχει μείνει ούτε ψίχουλο για τους υπόλοιπους, μόνο για τους ολιγάρχες. Λοιπόν, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε, εάν δεν αγγίξουν το διεφθαρμένο ολιγαρχικό ε, εκφυλισμένο σύστημα της ολιγαρχίας της Αρμενίας δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Πέστε μου λοιπόν τι λύση υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, θα ήθελα να αφαιρθώ στον Αγκορνό Καραμπάχα. Η σύγκρουση του Αγκορνό Καραμπάχα θα ήθελα να μου πείτε ε, κατά πόσον εσείς δεν θεωρείτε ότι είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο κουτί της Πανδώρας, διότι καταφέρετε να αναμίξετε με α, απίθανο τρόπο την εδαφική κυριαρχία που είναι η αρχή του Ελσίνκη ε, και ε, το Αζερμπαϊτζάν ε, ουσιαστικά λέει ότι είναι τμήμα της Αρμενίας και με τη συμφωνία Μαδρίτης Μης και τελικά δίνουμε το λόγο στους κατοίκους του από Καραμπάχα που σημαίνει ότι ε, ε, έχουμε εδώ το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Αν λάβουμε υπόψη μας λοιπόν ότι η συνέλευση του Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν θέλησε να ενταχθεί στο Αζερβαϊτζάν όταν το Αζερβαϊτζάν ανακήρυξε την ανεξαρτησία τους και όταν η αυτόνομη περιοχή της Νότιας Ισοτίας δεν χρειάστηκε, δεν θέλησε να ενταχθεί στη Γεωργία αντίστοιχα. Εάν αυτά τα δύο είναι ταυτόσημα δεν θα πρέπει να ακολουθούμε τα ίδια κριτήρια. Έχουμε τελείως διαφορετικά και το κουτί της Πανδώρας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας εφαρμόζεται πλήρως την κατάσταση στην Οσετία και έχουμε τελείως διαφορετικό κουτί της Πανδώρας ε, στην Κρυμαία. Για να λυθεί λοιπόν το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ ουσιαστικά αναφερόμαστε στη βούληση του λαού και το πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν τα πράγματα στην Κρυμαία. Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κουτί της στο οποίο έχουμε αλλάξει ε, το πολιτικό με το στρατηγικό όλο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Βενάρτ. Ε, εισηγούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα ε, λίγο μετά τις 5.30 διότι μετά έχουμε το νέο διοριστέντα επικεφαλή της αντιπροσωπείας για το Ισραήλ που θα μας συστηθεί εδώ, άρα έχετε περίπου πέντε λεπτά ο καθένας από τους προσκεκλημένους ομιλητές. Θα ξεκινήσουμε από τις κυρίες. Η κυρία Λίεβα, θέλετε να ξεκινήσετε για πέντε λεπτά και να απαντήσετε ορισμένες ερωτήσεις. Μετά η κυρία Μιναζιάν και στο τέλος ο κύριος Σούμπελ. Πέντε λεπτά ο κάθε ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματι, νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ και ε, δεν έχει δοθεί επαρκής προσοχή στο θέμα που είναι τόσο σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει πιο ε, έντονη εμπλοκή, πιο δραστηρία εμπλοκή, διότι είναι ένα θέμα που κρατάει την επιρροή της Ρωσίας στην περιοχή, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ισχύ, διότι υπάρχει επίσης και ένα θέμα εξοπλισμού που δεν μπορεί να τον, το αναχαιτήσουμε αυτή τη στιγμή και τα συμβαλόμενα μέρη ε, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όσο πιο πολύ στρατιωτικό πλεονέκτημα έχουν, τόσο πιο μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ αποκτούν δεν παραβλέπονται τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, δεν αποτελούν βάση για τις διαπραγματεύσεις, που είναι πολύ λυπηρό και εξηγεί γιατί η σύγκρουση συνεχίζεται και γιατί δεν ε, έχει σταματήσει. Υπάρχει μια ανασφάλεια και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε στη διαδικασία, μπορείτε να εμπλακείτε πιο ενεργά. Δηλαδή, μπορείτε να ε, δώσετε κάποιους προσανατολισμούς κανονιστικούς για τα δύο μέρη. Το άλλο θέμα είναι ότι η κοινωνία των πολιτών επικοινωνεί. Επικοινωνεί από την αρχή της διαδικασίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι στην Αρμενία έχουμε ανθρώπους που θέλουν, βλέπουν προς το μέλλον και εάν ε, δείτε τη μελλοντική προοπτική των χωρών. Η μελλοντική προοπτική έχει να κάνει με την συνύπαρξη, την ε, ενσωμάτωση, γιατί οι κοινωνίες και των δύο χωρών θέλουν να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε για... Ε, το, μιλάμε εδώ για τις κοινωνίες και το θέμα των απειλών είναι σημαντικό. Εξαρτώνται όμως από την πολιτική κατάσταση της χώρας και βλέπουμε πώς η ασφάλεια, τα πολιτικά θέματα, ο δημοκρατισμός είναι αλληλένδετα θέματα, διότι όσο πιο πολύ επηρεάζει η Ρωσία και ενισχύει την κατάσταση, τόσο πιο λίγες ε, δυνατότητες και ευκαιρίες έχουμε ε, για να κτίσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και αυτό έχει να κάνει και με την ε, ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Λίεβα. Τώρα η κυρία Μινασιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις και για τα σχόλια. Πραγματικά προτεραιότητα έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η χρηστή διοίκηση σε αυτή τη συμφωνία. Διότι αυτό υπερασπίζουμε από την αρχή και θέτουμε έμφαση στη σημασία αυτών των θεμάτων και για τις δύο χώρες, αλλά μπορώ να μιλήσω ιδιαίτερα για την Αρμενία. Αλλά είναι σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι η μόνη διασφάλιση της λογοδοσίας των εταίρων. Θα ήθελα να πω όμως ότι δεν είμαι ειδική σε θέματα γεωπολιτικής και ειρήνης. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω ότι η παρακολούθηση της ανακοχής και της κατάπασης του πυρός είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο δεν κατέστη δυνατόν. είναι τότε ένα τεράστιο εμπόδιο. Εμπόδιο στην πρόοδο της χώρας, της ειρηνικής ζωής στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν, αλλά και της οικονομικής, κοινωνικής πρόοδου και της δημοκρατικής ε, ανάπτυξης και των δύο χωρών, διότι είναι όμοιροι ε, στις συγκρούσεις αυτές και οι δύο χώρες είναι όμοιροι των καταστάσεων υπήρχε μια ερώτηση, αν κατάλαβα σωστά, για το ποια είναι η πολιτική βούληση ή οι πιθανότητες για σύναψη αυτής της συμφωνίας. Δεν έχω τη δύναμη να προβλέψω φυσικά, αλλά πιστεύω ότι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα οπισθοδρομήσουμε και δεν θα έχουμε αρνητική έκβαση. Ε, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία της χώρας. Από τη στιγμή που πρέπει να ε, προβεί σε μεταρρυθμίσεις και οι μεταρρυθμίσεις είναι κρίσιμη σημασία στην οικονομία, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πώς υλοποιεί η χώρα αυτά τα θέματα. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω. Αυτό αποτελεί τη μόνη εγγύηση ε, της πολιτικής βούλησης. Εάν η ελίτ, εάν τα καθεστώτα είναι έτοιμα να κάνουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ε, τότε γίνονται ελέγχοι στην εξουσία και οι μεταρρυθμίσεις, εάν ακολουθηθούν, τότε έχουμε κάποια ελπίδα ότι θα υπάρχει πολιτική βούληση και ότι θα υπάρχει πιθανότητα όντως να υπάρξει ανάπτυξη που θα αναχαιρετήσει την διαφθορά στη χώρα, θα βοηθήσει ε, τη χώρα και οικονομικά και κοινωνικά και από πλευράς ασφάλειας. Γι' αυτό ελπίζω ότι ε, οι προτεραιότητες είναι η χρηστή διοίκηση και τα ανθρωπινά δικαιώματα. Έγινε μια δήλωση ότι η Αρμενία έχει μόνο ένα φύλλο με αναφορά. Θα, πρέπει να σας βεβαιώσω ότι δεν αληθεύει, δεν ε, είναι μόνο ε, ο πρόεδρος της Αρμενίας, ο Ζέρ η Αρμενία συνεχίζει να βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως φίλο, ως ε, μια οντότητα που μπορεί να παραδώσει δικαιοσύνη. Και στρέφουμε ε, την προσοχή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρο. Διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρξε μια ερώτηση για το πώς βλέπουμε αυτό το θέμα. Νομίζω δεν, δεν έχω κάτι να προσθέσω για το πώς, τι είχε επιτευχθεί από αυτό τον διάλογο ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά και είναι αποτελεσματικός. Ε, γνωρίζω ότι η δυνατότητά μας να συμβάλλουμε στον διάλογο αυτό ε, είναι σημαντική και καταφέραμε να συμβάλλουμε στην, ε, στην πάταξη των γυναικής βίας, της, ε, ε, και καλωσορίζω αυτή τη δυνατότητα και υποστηρίζω το ότι η η διπλωματική γλώσσα δεν αναφέρεται στο να επιβάλλουμε, μα δεν μιλάμε για επιβολή, μιλάμε ε, για τη, την διαπραγματευτική μας θέση. Εάν απαιτούμε λογοδοσία, αν ζη... αυτό δημιουργεί την πολιτική βούληση και τη βάση δεν μιλάμε για επιβολή. Το πώς, ποια είναι η δυνατότητα των, της κοινωνίας των πολιτών, ποιες είναι οι δυνατότητές τους να κάνουν κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση. Με όλο το σεβασμό δεν έχω πολλές ελπίδες εδώ, διότι αυτή τη στιγμή και εδώ και αρκετό καιρό δυστυχώς βέβαια δεν είναι η τη λέξη, αλλά θα, θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για την αποτυχία της κοινωνίας των πολιτών, αλλά είναι ε, κυρίως η πολιτική κατάσταση στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν που δεν υποστηρίζει την κοινωνία των πολιτών στη συμμετοχή στο διάλογο. Προσπαθούμε Προσπαθήσαμε πριν από 10 χρόνια να ε, μπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών και ξέρω ότι έχει εμπλακεί σε διάφορα θέματα στην παρακολούθηση ε, του της έκφρασης λόγου. Τώρα είναι όλο ένα και λιγότερο δυνατό να εμπλακεί, όχι κατά ανάγκη λόγω της σύγκρουσης, μετά τον ε, περσινό πόλεμο των τεσσάρων ημερών είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά και χωρίς ε, ε, σύγκρουση οι δυνατότητες του, της κοινωνίας των πολιτών σε αυτό το διάλογο έχουν υποσκαφθεί σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, η πάταξη της ολιγαρχίας, υπάρχουν θέματα κατά της καταπολέμησης της ε, διαφθοράς. Όλα αυτά στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερικανική κυβέρνηση και στηρίζονται επίσης ε, με εμπειρογνώμονες και πόρους και είναι σημαντικό αυτή η καταπολέμηση να φτάσει ε, να γίνει όσο πιο έντονη, διότι αλλιώς θα παγιδευτούμε σε αυτό τον αέναο αγώνα χωρίς να έχουμε πραγματικά περιορισμό της ε, εξουσίας. Ευχαριστώ. And finally, Mr. Schubel. Ευχαριστώ κύριο Σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Κύριε Τάνοκ και κύριε Νικολάη, προφανώς οι τελευταίες εξελίξεις, η κλιμάκωση έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, μόνο ειρηνική. Πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό, καθώς οι στρατιωτικές δραστηριότητες οδηγούν μόνο σε αδιέξοδο. Κατόπιν ε, θεωρώ ότι οι ε, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μας δώσουν πολύ περισσότερες δυνατότητες και συνεργασία με τις νέες συμφωνίες για να συζητήσουμε για το κράτος δικαίου. Έχουμε έναν ε, ειδικό απεσταλμένο, τον κύριο Ζάλπερ για τον Νότιο Κάφκασο και θα τον διαδεχτεί κάποιος, δεν έχει ακόμα επιλεγεί είναι βεβαίως συμπρόεδρος στην ομάδα του Μίνσκ και συνεργάζεται στενά προφανώς με τους Γάλλους ε, συναδέλφους. Πράγματι τα αποτελέσματα της ομάδας του Μίνσκ δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά όσο θα θέλαμε δηλαδή να επιληθεί η σύγκρουση, αλλά ίσως η ύπαρξη της ομάδας αυτής απέτρεψε τα χειρότερα. Μια κλιμάκωση. Νομίζω ότι αυτό είναι από μόνο του ένα επίτευγμα. Αν δούμε Βεβαίω στην τελευταία κλιμάκωση ίσως όχι και τόσο εντυπωσιακό. Κύριε Γκάλερ, για την Αρμενία. Είχαμε την εντύπωση πρώτα απ' όλα όταν διαπραγματευτήκαμε την Συμφωνία Σύνδεσης με την Αρμενία μέχρι το 2013 ότι η Αρμενία είχε εμπλακεί πλήρως και η Αρμενία χρειάστηκε τις συντομότερες διαπραγματεύσεις λιγότερο και από την Γεωργία και τη Μολδαβία τελικά βεβαίως δεν στέφθηκε με την σύναψη της συμφωνίας που θα θέλαμε. Τώρα δεν θέλω εγώ να κάνω εικασίες για τους λόγους. Η νέα συμφωνία μετά από την περίοδο αυτήν περισυλλογής είχαμε και έχουμε την εντύπωση ότι η Αρμενία θέλει να λειτουργήσει και η νέα αυτή συμφωνία και νομίζω ότι Έχουμε κάποιους μοχλούς πίεσης και ήμασταν ιδιαίτερο επιτυχημένοι όταν, παραδείγματο χάρη, καταφέραμε να έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα στις τελευταίες εκλογές. Και εδώ πέρα δείχνουμε ακριβώς ε, το πώς μπορεί να λειτουργήσει η στήριξη της Ένωσης. Βεβαίως η δήλωσή μας λέει ότι δεν ήταν τέλεια τα πράγματα, αλλά ήταν παρόλα αυτά κάτι το θετικό. Με τη νέα συμφωνία λοιπόν θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες να συνεργαστούμε στενότερα με την αρμενική πλευρά. Το ίδιο και για το Αζερβαϊτζάν βεβαίως. Κύριε Βάγγελ, ναι, συμφωνώ. Πρέπει να βρεθεί μια λύση με βάση το διεθνές δίκαιο, αυτό είναι σαφές. Και ο ρώτησε για την ένταξη του Αζερβαϊτζάν στον ΠΟΕ ε, ίσως χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμα. Το Αζερβαϊτζάν δεν είχε εμπλακεί σε διαπραγματεύσει με τον ΠΟΕ εδώ και καιρό. Τώρα υπάρχει κάπως μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί θέλει να αναπτύξει ποικίλο τρόπο στην οικονομία του. Μα η αίσθησή μου είναι ότι ίσως μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαπραγματεύσεις γιατί χρειάζονται και διμερείς συμφωνίες με τα μέλη που το επιθυμούν Οπότε καλό είναι να προχωρήσει η δικιά μας η συμφωνία, η οποία έχει εμπορικό σκέλος, απλά δεν μπορεί να είναι τόσο φιλόδοξο όσο θα ήταν. Για την Ευρασιατική Ένωση, το ανέφερε και ο κ. Σαστοβίτσιουτς, προφανώς ε, δεν είμαστε σε επίσημο διάλογο με την Ευρασιατική Ένωση. Ε, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αν μιλήσετε σε ε, μεμονωμένα κράτη-μέλη της Ένωση, Ένωσης ε, θα έχετε κάποια ιδέα, αλλά όπω σα είπα δεν έχουμε κάποια επίσημη σχέση και αυτή δεν επηρέασε καθόλου με τη σειρά τη και τη συμφωνία μας. Πρέπει βεβαίω να λάβουμε υπόψη, η Γερμανία μάλλον, το τι θέλει να συμφωνήσει μαζί μας. Βεβαίως σαφές είναι ότι καμία άλλη ένταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει την διμερή μας συμφωνία. Η δημιουργή μας συμφωνία προηγείται. Η συμμετοχή σε καμία άλλη λέσχη δεν μπορεί να προηγηθεί. Τώρα, από τον Ισπανό βουλευτή ότι ελέγχουν οι ολιγάρχες στην χώρα. Ε, αυτό δεν είναι καινούριο, ούτε αφορά μόνο την ε, Αρμενία. Είναι γενικό στον μετασοβιετικό χώρο το φαινόμενο. Και νομίζω ότι με το κράτος δικαίου, με νέες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταφέρουμε να μοιέσουμε ακριβώς ε, την επιρροή αυτή. Και η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι όρος εκ των όνων μας και από αυτού συνεργαζόμαστε και με την Αρμενία και με τις άλλες χώρες της Ανατολική Γειτονία. Για τον Αγκόρνο Καραμπάχ και το κουτί τη Πανδώρας. Όλες οι συγκρούσεις στην περιοχή είναι πολύ επικίνδυνε. Πολλοί λένε ότι είναι περίπλοκο τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Όλες αυτές οι συγκρούσεις είναι επικίνδυνες και εμποδίζουν και την ανάπτυξη. Αν δείτε τι οικονομικές δυνατότητες ε, θα είχαν η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν από αυτή τη σύγκρουση. Νομίζω και εσείς θα θέλατε να τελειώσει αυτή η σύγκρουση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας, ε, την κυρία Λίεβα, την κυρία Νασιάν και τον κύριο Σούμπολ που μπήκαν στο χρόνο να μας απαντήσουν. Πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο, θα ήθελα να πω δύο λόγια ε, λόγω και των προσφάτων γεγονότων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Επειδή έχουμε πολύ δραστήριους συναδέλφους που ασχολούνται και με το Αζερβαϊτζάν και με την Αρμενία, ε, που όμως δημοσίευσαν τελείως διαφορετικά ανακοινοθέντα στον τύπο τις τελευταίες ημέρες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Καρίμ πρόεδρος της ε, ε, αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Αζερβαϊτζάν, ε, η κυρία Χάρμς ως πρόεδρος του Λιούρανου και εγώ ως πρόεδρος της ΑΦΕΤ, κάναμε την εξή κοινή δήλωση στις 6 Ιουλίου που καλύπτει την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα για την ανανέωση της βίας ε, την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν που οδήγησε και πάλι στο θάνατο αμάχων στην περιοχή του Φιζούλη. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, ζητάμε άμεση διακοπή των εχθροπραξιών μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν και όπως είπαμε προηγουμένως πιστεύουμε ότι η σύγκρουση Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν έχει στρατιωτική λύση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, μια πολιτική επίλυση βάσει διεθνή δικαίου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει η περιττή ε, ε, αυτή η κατάσταση των θανάτων αμάχων και στρατιωτών από τις δύο πλευρές. Υποστηρίζουμε τις διαδικασίες διαμεσολάβησης και τις προτάσεις της ομάδας ε, του ΜΙΣΚ ε, και για να υπάρξει αυτή η διαμεσολάβηση και η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν πρέπει να βρουν το πολιτικό στένος να διαπραγματευτούν καλή την πίστη. Αυτή είναι η δήλωση και ελπίζουμε να μπορέσει να υπάρξει μια λύση. Ε, περνάμε στο επόμενο σημείο, το παρεθμό 6. Να θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι αυτό το σημείο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, επομένως μόνο τα μέλη, ε, εγκεκριμένε πολιτικές ομάδες και προσωπικό να παραμείνουν. Σας παρακαλώ όλοι οι υπόλοιποι να απαχωρήσουν.